Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να καθίσουμε όσοι έχουν έρθει για την ακρόαση και να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Καταρχήν το σημείο 1. Θα σας υποβάλω κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Τα σημεία 6 και 7 για την πορεία των διοργανικών διαπραγματεύσεων για την μπλε κάρτα και τον ε, κανονισμό για τις δεξιότητες αναβάλλονται για, την, για μια επόμενη μας συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσει αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη, την εγκρίνουμε με αυτές τις αλλαγές. Καταργή, ε, για τη διερμηνία, να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε διερμηνία στα μαλτέζικα, κροατικά και γοεδελικά. Έγκριση των αποφάσεων, των συστάσεων των συντονιστών. Διορισμός ηγητών. Καταρχήν η κυρία Ζίπελ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, ανέλαβε την έκθεση ε, για την πρόταση κανονισμού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το σεβασμό της ε, προσωπικής ζωής και την προστασία προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Όσοι έρχονται κάπως καθυστερημένα για τη συνεδρίασή μας, έχω ξεκινήσει ήδη τη συνεδρία τη Επιτροπή, γι' αυτό παρακαλώ καθίστε αθόρυβα. Κανονικά πρέπει να είμαστε στην ώρα μα. Λοιπόν, η κυρία Ζήπελ ανέλαβε την ε, έκθεση τη πρόταση κανονισμού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το σεβασμό τη ε, προσωπική ζωή και την προστασία προσωπικών δεδομένων στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Η κυρία Κουντρίτσκα είναι του ΕΛΚΑ επίση. Ε, εισηγήτρια γνωμοδότηση τη έκθεση πρωτοβουλία Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για την ε, ετήσια έκθεση του 2016 και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Ε, συμφωνούμε να εγκρίνεται. Επίση, ε, κατά εξοδότηση πράξη, έχουμε λάβει στι 28 Οκτωβρίου ένα σχέδιο εκτελεστική απόφαση ε, για την αυτοματοποιημένη αναταλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά την καταγραφή των οχημάτων στην Πορτογαλία. βασική πρόταση, απόφαση για την καταπολέμηση της του διασυνοριακού εγκλήματος. Ε, η λήψη αυτής της εκτελεστικής πράξης έχει, θα μοιραστεί μέσα της, ε, του εντύπου ενημερωτικού της ε, Επιτροπολογής 8 Δεκεμβρίου 2017 και ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν να επιληφθεί. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες ακριβώς στις 11 Οπότε να είστε έτοιμοι για τις 11, να έχετε έτοιμες ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Έγκριση πρακτικών 24-25 Απριλίου και 29 Ιουνίου 2017. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και περνάμε τώρα στο πρώτο κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η ακρόασή μας για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι. σα καλωσορίζω θερμά σε αυτή τη δημόσια κρόση για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Και πάλι να σα πω ότι δυστυχώ δεν έχουμε διερμηνία στα μαλτέζικα, κροατικά, κοδελικά, αλλά έχουμε σε όλε τι υπόλοιπε γλώσσε. Επίση, ε, μεταδίδεται απευθεία στο διαδίκτυο η δημόσια κρόση. Και επίση, οι συντονιστέ αποφάσισαν στη συνεδρίαση τη 24η Οκτωβρίου 2017 την οργάνωση δημόσια κρόαση ε, ως προπαρασκευαστικό έργο της ειδική έκθεσης που με βάση το άρθρο 83 του ιστορικού κανονισμού θα εκπονήσουμε για την κατάσταση στην Ουγγαρία όπως προέβλεψε το ψήφισμα της Ολομέλης της 17ης Μαΐου 2017. Στη συνεδρίαση της 13 η Νοεμβρίου 2017 το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε έγκριση για την διοργάνωση δημόσιας ακρόασης στις 7 Δεκεμβρίου και με επιστολή τη 23 η Νοεμβρίου ο πρόεδρο Σταγιάννη με ενημέρωσε για την απόφαση του Προεδρείου. Να επισημάνω ότι 21 Νοεμβρίου οι συντονιστέ τη Επιτροπής μας αποφάσισαν για τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κατάλογος αυτός περιλάμβανε και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής της Βενετίας αλλά μια και συμπίπτει η συνεδρίασή μας με την 113η συνεδρίαση 8 και 9 Δεκεμβρίου της Υποεπιτροπής ε, στη Βενετία. Δυστυχώς εκπρόσωπος της Επιτροπής της Βενετίας που είναι του, Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατία μέσω του δικαίου αδυνατεί να παραστεί. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ε, έδωσα άδεια στο κανάλι της Ουγγρικής Δημόσιας Τηλεόρασης να μαγνητοσκοπήσει τη συνεδρίασή μας. Επειδή έχουμε μόνο δύο ώρες για τη δημόσια ακρόαση και όπως είπα η ακρόαση είναι πολύ σημαντική, θα φροντίσω να τηρηθεί ευλαβικά ο χρόνος αγόρευσης και το λέω αυτό προς γνώση και συμμόρφωση όλων των ομιλητών. Πριν να σας δώσω το λόγο θα σας ενημερώνω για το χρόνο που δικαιούστε. Θα δώσω πρώτα όμως το λόγο στην εισηγητριά μας για το θέμα της Ουγγαρίας που είναι η κυρία Γιουντίτ Σαρχεντίνη. Εσύ, Γιουντίτ, έχεις 10 λεπτά. Πολύ γενναιόδωρο από μέρου σου. Δεν νομίζω θα εξαντλήσω το δεκάλεπτο, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά και ένα θερμό καλώς όρισμα θα ήθελα να απαθήνω στους καλεσμένους μας και πριν να ακούσουμε τις δικές τους δηλώσεις θα ήθελα να σα ενημερώσω για το σκοπό αυτή τη δημόσια ακρόαση και το εγχείρημα Γενικώ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Φέτο το Μάιο το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή μα ε, την έναρξη τη διαδικασία και την εκπόνηση ειδική έκθεση προκειμένου να ψηφιστεί στην Ολομέλεια η πρόσφατη πρόταση του, του Συμβουλίου ε, για την εφαρμογή του άρθρου 7.1 της Εθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το άρθρο 83 του εσωτερικού μας κανονισμού. Ε, και μάλιστα το Κοινοβούλιο έλαβε αυτήν την απόφαση γιατί όπως αναφέρεται στο ψήφισμά μας ε, θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά εμφανή κίνδυνο σοβαρή κατάφορης παραβίασης των ε, αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της συνθήκης. Οπότε εγκαινιάζει την ε, διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1. Επίσης, ε, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι εξελίξεις στην Ουγγαρία οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων της ελευθερίας έκφρασης, ε, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ανθρώπινα δικαιώματα των, των άσυλων, των μεταναστών προσφύγων, δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, παρακόλληση των ε, δραστηριοτήτων ε, των οργανώσεων κοινωνία πολιτών, δικαίωμα τη μεταχείριση, δικαιώματα μειονοτήτων, των, μεταξύ άλλων Ρωμά, Εβραίων, LGBTI, ε, παραβίαση κοινωνικών δικαιωμάτων, παρακόλληση λειτουργία του θεσμικού συστήματο, ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία και άλλων θεσμικών φορέων και έχουμε και πολύ ανησυχητικέ καταγγελίε για σύγκρουση συμφερόντων και διαφθορά. Όλα αυτά μαζί ε, συνιστούν ένα συστημικό κίνδυνο ως προς το κράτος δικαίου μιας χώρας μέλος. Επίσης θεωρούμε ότι η Ουγγαρία είναι η λιδία λίθος για να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ετοιμότητα και την ικανότητά της να αντιδράσει σε απειλές ή παραβιάσεις των θεμελιωδών της αξιών από κάποιο κράτος μέλος. Και με ανησυχία επισήμανε ότι εξελίξει και σε άλλα κράτη-μέλη δείχνουν επίσης ανησυχητικά σημάδια υπονόμευση του κράτους δικαίου αντίστοιχα με αυτά τη ουγγαρία. Επίσης, το Κοινοβούλιο έκρινε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος και ότι θα πρέπει το έργο μας να ολοκληρωθεί με μια αμερόληπτη ε, συνεργασία και με μια, μετά από μια συνεργατική διαδικασία. Επίσης, έχουμε την ανακοίνωση του 2003 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 7 τη συνθήκη που προβλέπει ε, σεβασμό και προαγωγή των ιδρυτικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Στην ανακοίνωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 7 δεν περιορίζεται στους τομείς του ενωσιακού δικαίου. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δρά όχι μόνο σε περίπτωση παραβίασης των κοινών αξιών σε περιορισμένους τομείς, αλλά ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης σε ένα τομέα όπου το κράτος έχει αυτόνομη δράση. Επίση, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το άρθρο 7 δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίωμα δράση, που είναι πολύ διαφορετικό από τι ε, εξουσίε τη της ε, στήριξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη απέτηση να το κάνουν τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Οπότε το ψήφισμα του Μαΐου και με βάση και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2003 είναι οι βάσεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την εκπόνηση της έκθεσής μου. Και μάλιστα αυτή η δημόσια ακρόαση είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης στοιχείων. Γι' αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τις ε, ομιλίες σας, γιατί όλες οι γνώσεις που θα συγκεντρώσουμε σήμερα θα συμπεριληφθούν στην έκθεσή μου, το σχέδιο της οποίας θα υποβληθεί το Μάρτιο. Ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη, ήσασταν η συγγήτρια θα δώσω τώρα το λόγο καταρχάς στον Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας ε, για 10 έως 12 λεπτά. Eh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σάρατο. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμε ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω τα ζητήματα αυτά ενώπιον της Επιτροπής σας και να σας ενημερώσω για την θέση της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Πραγματικά σας ευχαριστώ για την προσοχή που συνεχίζετε να προσδίδετε στην ε, κατάσταση και στις εξελίξεις στη χώρα με την Ουγγαρία και είναι πολύ θετική αυτή η δυνατότητα να συζητήσουμε την κατάσταση γιατί οι Ούγγροι ε, θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αντιπαραβολή απόψεων, ε, συζήτηση, διάλογος. Ε, άλλωστε πρόκειται για τα θεμέλια της δημοκρατίας. Μας αρέσει ο διάλογος, ποτέ δεν αποφεύγουμε λοιπόν το διάλογο. Ακόμη και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει αντιπαραθέσεις. Και ένας άλλωστε από τους λόγους που προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και άλλωστε θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακριβώς η δυνατότητα να συζητήσουμε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και να επιλύσουμε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Νομίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους και να τις υπερασπιστούν. Επομένως, είναι αντιδημοκρατικό και αντιβαίνει στις αξίες της Ένωσης εάν κάποιος αρνηθεί το δικαίωμα μιας χώρας να προασπίσεται τις θέσεις της ή της ερμηνείας των ζητημάτων που την αφορούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις ε, στην Ουγγαρία. Ταυτόχρονα και εμείς παρομοίως παρακολουθούμε και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ισχύει και τη δική σας επιτροπή. Πρέπει να πω ότι σε πολλά θέματα ε, αντιλαμβανόμαστε εντελώ διαφορετικά την έννοια έθνος, εθνική υπερηφάνεια, σεβασμός παραδόσεων, προσέγγιση στη θρησκεία, ασφάλεια, διαχείριση συνόρων. Φαίνεται να είμαστε σε διαμετρικά αντίθετες ε, θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι δεν θα σας αρέσουν και πολύ αυτά που θα σας πω. Πάντως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στους Ούκρους δεν αρέσουν και πολύ κάποια πράγματα που λέτε εσείς εδώ, ούτε ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεστε στη χώρα μας. Διότι πράγματι επιτίθεστε στη χώρα μας, αγαπητοί βουλευτές. Άρα έρχεστε αντιμέτωποι με αυτόν τον τρόπο, με μια χώρα η οποία την ισχύ της, ε, την αντλή, από το να δημιουργεί λύσεις από προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια η Ουγγαρία έκανε πάντα δυνατόν, ώστε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε πάντα δυνατόν, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανακτήσει έστω και ένα μέρος της απολεστής ανταγωνιστικότητάς της. Η οικονομική μας κατάσταση ήταν αρχικά χειρότερη ακόμη και από της Ελλάδας και μας κρατούσε ε, ζωντανό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχαμε πάνω από 85% ε, έλλειμμα Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή όμως αρχίσαμε ένα νέο πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αμφισβητήθηκε από πολλούς. Πάντως αποκαταστήσαμε την ε, ισορροπία στον προϋπολογισμό ένωσαν τις δυνάμεις τους ε, οι Ούγγροι, αναγνώρισαν το έργο μας ε, και είδαν επίσης ότι όλα τα προβλήματα, ακόμη και τα πιο δύσκολα, μπορούν να επιληθούν. Έχουμε 750.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε έλλειμμα κάτω του 3%. Έχουν ξεκινήσει νέες ε, επαγγελματικέ στατιοδρομίε. και έχουμε τους χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης της απασχόλησης. Μας αρέσει να είμαστε ντόμπροι στις ε, κουβέντες που λέμε. Να λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Η πολιτική ορθότητα πραγματικά έχει συγκαλύψει πλέον την ειλικρίνεια του διαλόγου. Άρα νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ο ένας με τον άλλο, να συζητάμε τα πράγματα ανοιχτά. Και αν το κάνουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους, που έχει να κάνει και με το πεπρωμένο της Ευρώπης, αν θέλετε. Λαφρομετανάστευση. μετανάστευση. Η Ουγγαρία αντιλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίπτουμε την λαθρομετανάστευση και τις τεχνητός οριστήσεις ποσοστώσεις. Θεωρούμε ότι η λαθρομετανάστευση αποτελεί μια σοβαρή απειλή. Το αποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές εξελίξεις τα δύο τελευταία χρόνια. 1,5 εκατομμύριο είναι οι λαθρομετανάστες που έχουν έρθει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εντελώς ανεξέλεγκτα, φτάνουν στα σύνορα επιτίθενται στους αστυνομικούς, παραγνωρίζουν τους νόμους μας, δεν σέβονται την, ε, ε, τις συνήθειές μας, τον τρόπο ζωής μας. Έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις με πάνω από 330 νεκρούς και πάνω από 1.200 τραυματίες η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει. Αυτό όμως η Ευρώπη δεν θέλει να το ε, αποδεχθεί. Δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι πρέπει να ζούμε υπό το φόβο της συνεχούς τρομοκρατικής απειλής. Πρέπει λοιπόν για μας να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορα της Ευρώπης. Και εμείς οι Ούγγροι θεωρούμε ότι στην Ευρώπη η ασφάλεια πρέπει να ενισχυθεί και να αποκατασταθεί. Μέχρι στιγμής δαπανούμε 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το δικό μας μερίδιο το δικό μας λιθαράκι στην προσπάθεια προστασίας ε, των εξωτερικών συνόρων της Ένωση, των συνόρων του Σέγγεν. Για να τηρήσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόσφατα λάβατε στην Επιτροπή σα αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μια απόφαση η οποία σημαίνει ουσιαστικά υποχρεωτικό μηχανισμό ε, μετεγκατάστασης με κάποιες εξελίξεις ε, που ανεπιστρεπτή θα οδηγήσουν στη μόνιμη και ανεφόρον ε, μεταγκατάσταση όπως είπε κάποιος, ενός εκατομμυρίου ε, ο ε, παράνομων ε, μεταναστών. Το σύστημα όμως αυτό έτσι θα καταρρεύσει, αυτό είπε ο Τζορ Σόρος. Και αυτό σχετίζεται σίγουρα και με την απόφαση αυτή. Τέτοιου είδου αποφάσει είναι επικίνδυνε γιατί μπορεί να πείσουν ε, μάζε ολόκληρε ε, ανθρώπων να φύγουν από του και να προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και έτσι να υποβαθμιστεί η ασφάλεια μια χώρα αλλά και να ε, τη στερηθεί η δυνατότητα να αποφασίζει ποιο θέλει να έρθει στη χώρα τη και με ποιον θέλει να συμβιώνει στη χώρα της. Μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αποφάσεις, να τις πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Όπως βεβαιώνουν και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν τα ζητήματα αυτά εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς οι Ουγγροί στρεφόμεθα για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του έθνους μας, ε, τους πολίτες της χώρας μας. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών, εσείς οι βουλευτές, δεν ζητάτε τη γνώμη των ε, Ευρωπαίων πολιτών με εθνικούς μηχανισμούς διαβούλευσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί πρέπει οι πολίτες να δίνουν την απόψη τους για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Έχουν αυτό το δικαίωμα και είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να το κάνουν εφόσον θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν το λαό τη χώρα του. Η Ουγγρική κυβέρνηση, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, φυσικά και ζήτησε την άποψη των Ούγγρων πολιτών για το θέμα τη παράνομη μετανάστευση. Δεν ξέρω πώ από εσά ε, κατάγεστε από μια χώρα που υπήρξε διαβούλευση, υπάρχουν διαβουλευσει ε, με του πολίτε για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο να μπορείτε να βασίζεστε και μια σαφή άποψη των πολιτών για αυτά τα θέματα. Στην Ουγγαρία, τρία εκατομμύρια πολίτε ε, τάχθηκαν κατά τη μετανάστευση ε, και στο πλαίσιο τη Εθνική Διαβούλευση ε, συμμετείχαν δύο εκατομμύρια άνθρωποι που έδωσαν τι απόψει και είπαν όχι στην παραμετανάστευση. Είπαν όχι στι υποχρεωτικέ ποσοστώσει αναδεκατάσταση. Η Ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει παρά να εκπροσωπήσει τη βούληση του γκρικού λαού και να προσπαθήσει να εφαρμόσει στην πράξη τη βούληση αυτή. Εμείς προσπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ούγγρων πολιτών, την ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και της χώρας. Πιστέψτε με, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, θα αναλώσουμε κάθε εκμάδα για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε απόφαση στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της Ουγγαρίας. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στις συζητήσεις μας θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή την άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ που μας υποδεχθήκατε σήμερα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Η Ουγγρική Κυβέρνηση και στο μέλλον θα δείξει την ίδια ετοιμότητα να προασπίσει τις θέσεις της, τις θέσεις των Ούγγρων πολιτών. Νομίζω ότι στην Ευρώπη καλό είναι να υπάρχει διάλογος, καλό είναι να συζητούνται τα θέματα, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δημοκρατία. Σας ευχαριστώ και πάλι και για τη δυνατότητα και για την προσοχή που μου ε, δώσατε να μιλήσω και για την προσοχή που αποδίδεται στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Μάρτα Παρντάβη, ε, συμπρόεδρος ε, της Ουγγρικής Επιτροπής του Ελσίνκη. Έχετε και εσείς 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έρθω να μιλήσω εδώ σήμερα. Αποτελεί τιμή ε, ως εκπρόσωπος ε, μιας ε, ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συστήθηκε το 1989 στην Ουγγαρία. Ε, έχουμε ως στόχο να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία. Η Επιτροπή του Ελσίνκη επικεντρώνεται στην προστασία των προσφύγων, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτηση ε, και τήρηση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χαρήκαμε που ήμασταν ε, στον κατάλογο για το βραβείο Βάτσλακ Χάβελ και λάβαμε και ε, το βραβείο του Πορτογαλικού Ιδρύματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα και είναι πολύ δύσκολο για μένα σήμερα να να απαντήσω στα σχόλια του Υπουργού, ε, το οποίο θα γίνει αργότερα σήμερα, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν υποθεί καν. Πολύ σημαντικές ε, ανθρώπινες αξίες, οι οποίες δεν εκφράστηκαν στην προηγούμενη παρέμβαση και αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αυτές είναι κοινέ αξίες εγγεγραμμένες στο άρθρο 2 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν κοινέ αξίε που αποτελούν και του πυλώνε, αλλά και τους κοινωτήρους μοχλούς ε, τη Ευρωπαϊκή κοινότητα και τη Ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωσης. στην Ουγγαρία όμω είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ουγγρική κυβέρνηση αποδυναμώνει συνεχώς ε, του ελέγχου και τι δικλείδε ασφαλείας και τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Ε, υπάρχει συνεχής απειλή για τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν γίνονται σεβαστές συνεχώς σε μια χώρα όπου τα θεσμικά όργανα έχουν αποδυναμωθεί ή έχουν και διαλυθεί τελείως σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος της κοινωνίας των πολιτών για να μπορούμε να αντισταθμούσουμε την επιβολή αυτή της εξουσίας. Θα πρέπει το, ε, η κυβέρνηση να είναι υπόλογη και αυτό δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αν δεν υπάρχει πολυφωνία των μέσων, ελεύθερα μέσα και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών έχει πολλούς ρόλους, αλλά ένας είναι πάρα πολύ σημαντικός εδώ σήμερα και αυτό είναι να ε, λέμε την αλήθεια ενώπιον της εξουσίας. Ως οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουμε ανθρώπους, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της ε, για την κατάχρηση εξουσίας και την παραβίαση των ε, βασικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 2. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ακούγοντας την Ουγγρική κυβέρνηση ε, να προτάσει το επιχείρημα και να ισχυρίζεται ε, ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική τακτική, μια πολιτική τακτική την οποία εκμεταλλεύεται ο τύπος ή ε, θεωρείται παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα, ανάμιξη στις αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Αυτό που ακούω ουσιαστικά είναι ότι ε, η Ουγγρική κυβέρνηση αμφισβητεί την κοινή φύση των κοινών μας βασικών αξιών. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών όμως είναι να ενθαρρύνει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις και τους υπολείπους να δρούν προς το συμφέρον της τήρησης των βασικών μας αξιών. Η έκφραση των πολυφωνικών απόψεων στην Ουγγαρία ε, συρρυκνώνεται συνεχώς, ιδίως την τελευταία χρονιά. Και αυτό φυσικά καλύπτει ε, και μια πολύ επιθετική εκστρατεία προπαγάνδας που ξεκίνησε το 2013 κατά της κοινωνίας των πολιτών με συγκεκριμένα μέτρα για να χαθεί αξιοπιστία και να ε, φοβήσουν ανεξάρτητα με ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οργανώσεις που θέλουν να είναι υπόλογες κυβερνήσεις για τις παραβιάσεις και τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Θα θυμάστε βεβαίως ε, τη σειρά των χωρίς καμία αιτιολογία ερευνών που έγιναν, ακόμα και αστυνομικές έρευνες το Σεπτέμβριο του 2014 κατά μη κυβερνητικών οργανώσεων που είχαν ε, λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ορβηγία. Υπήρχαν και άλλα μέτρα τα οποία πίεζαν ε, την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και αυτό ε, περιλέμβανε και ισχυρισμούς χωρίς καμία απόδειξη από τις κυβερνήσεις, παραπλανητικές εκθέσεις ε, και από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και από μέσα τα οποία τάσσονται με την κυβέρνηση. Υπήρχαν εκστρατείες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος και θα θυμάστε ε, ότι υπάρχαν ε, πανό τα οποία ζητούσαν να σταματήσουν οι Βρυξέλλες, έκαναν επίθεση στα θεσμικά όργανα και υπάρχει και μια πρόσφατη συζήτηση η οποία φοβίζει τη χώρα με ένα σενάριο ε, καταστροφής λόγω της μετανάστευσης. Αυτά όλα είναι κατά ανθρώπων και ομάδων που εκφράζουν απόψεις για τα δημόσια θέματα τα οποία είναι αντίθετα με την Ουγγρική κυβέρνηση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σεβασμό των κοινών αξιών σε μια δημοκρατία. Ο ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήρθε στην Ουγγαρία και δημοσίευσε την έκθεσή του το Μάρτιο φέτο και εκεί εξέφρασε την ανησυχία του για το συνεχή στιγματισμό των ανθρώπων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται γλώσσα συγκεκριμένη από τις ε, κυβερνήσεις και από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και στο ψήφισμά του του Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ουγγρική κυβέρνηση, θα το θυμάστε, να αποσύρει την τότε πρόταση ε, νόμου για τους ε, οργανισμούς και οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά εγκρίθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ε, ε, και έχει γίνει γνωστός ε, ο νόμος κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και παγκοσμίω και βάσει αυτού του νόμου οποιαδήποτε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών λάβει πάνω από 23.000 ευρώ ξένης χρηματοδότησης πρέπει να εγγράφεται στα Μητρέο ως οργάνωση η οποία χρηματοδοτείται από το εξωτερικό. Η χρηματοδότηση μπορεί να έρχεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα Ηνωμένα Έθνη, από ιδιώτες, ε, Ούγγρους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό ή πολίτες οι οποίοι αποφασίζουν να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών στην Ουγγαρία από το εξωτερικό. Αυτή η ε, ξένη χρηματοδότηση πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα δημοσιεύματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε είναι έντυπα, ε, είτε είναι στο διαδίκτυο. Ε, εάν δεν τηρηθεί αυτό, μπορεί να υπάρχουν και πρόστιμα και μπορεί τα δικαστήρια να αποφασίσουν τη διάλυση του οργανισμού. Η ε, Επιτροπή ε, της Βενετίας εξέδεσε μια απόφαση ε, για το νομοσχέδιο αυτό μια εβδομάδα μετά την έγκρισή του και είπε ότι παρά τι καλέ προθέσει, ε, το νομοσχέδιο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να μαυρώσει την εικόνα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αντιβαίνει στην ελευθερία τη έκφραση, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση για το συγκεκριμένη νομοθεσία κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και σήμερα πολλέ ουγγρικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν εκφράσει δημοσίω την άποψη ότι ο νόμο αυτό είναι εντελώ περιττό σε μια δημοκρατική κοινωνία, στιγματίζει και είναι επιζήμιο. Και είναι απαραίτητο να γίνει αυτό διότι οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών ήδη είναι ιδιαίτερα διάφανε. Στιγματίζει διότι ε, οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται προ όφελο τη ουγγρική κοινωνία μέσω πόρων που μπορούν να συλλέξουν από το εξωτερικό θεωρείται ότι απειλούν τη χώρα. Και είναι επιζήμιο διότι υποδαβλίζει την ε, δημοκρατία, βυσβητεί το δικαίωμα της ελευθερίας και το δικαίωμα της έκφρασης και ε, υπάρχουν λόγοι να πιστεύετε ότι αυτή η πρόσφατη νομοθεσία δεν θα είναι ε, το τέλος αυτής της κυβερνητικής εκστρατείας κατά της κοινωνίας των πολιτών. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα σε μια μακρά διαδικασία και ε, ε, είναι αντίστοιχο με το μοντέλο που βλέπουμε στη Ρωσία και μάλιστα ομοιάζει πάρα πολύ ε, με τον νόμο για τη Ρωσία, για τους ξένους πράκτορες ε, που ουσιαστικά έχει στιγματίσει τους, ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη Ρωσία και η θέση τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα πολλές χρειάστηκε να κλείσουν στη Ρωσία. Και η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει πάρα πολλές ομοιότητες με την νομοθεσία της Ρωσίας. Εκστρατείες για να μαυρωθούν συγκεκριμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως αυτή για την οποία εργάζομαι ομοιάζει πάρα πολύ με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Ρωσία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τώρα τελευταία η κυβέρνηση άρχισε να αναφέρεται σε κινδύνους εθνικής ασφαλείας. Ήδη από τον Νοέμβριο ο Πρωθυπουργό και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης ανέφεραν ε, ότι έχουν δώσει οδηγίες στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας για να δουν πώς ε, έχει δει ε, σχέση το δίκτυο με τις Βρυξέλλες, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως ε, Ούγγρος πολίτης, εγώ προσωπικά ανησυχώ πολύ, διότι αντί να ε, βοηθά την ανοχή, η Ουγγρική κυβέρνηση ε, πυροδοτεί τη μυσαλλοδοξία και υπάρχουν καταχωρήσεις και πανό τα οποία είμαι βέβαιη ότι θα έχετε δει, τα κονδύλια τα οποία ε, δαπανώνται από την κυβέρνηση οδηγούν ε, σε μυσαλλοδοξία και σε ρατσισμό, ε, φόβο, ξενοφοβία κατά των μεταναστών και των προσφύγων, κυρίως κατά των μουσουλμάνων και αυτό έχει δημιουργήσει μίσος και φόβο στην κοινωνία. Σε πολύ μικρές κοινότητες δεν έχουν επιτραπεί κάποιοι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να κάνουν καν διακοπές στα χωριά τους και ξένοι που διαμένουν σε τοπικά ξενοδοχεία ή ε, ξενώνες χρειάστηκε να δείξουν επιστοποιητικά ότι έχουν εμβολιαστεί. Ε, τέτοιες ριζοσπαστικές, εξτρεμιστικές απόψεις, ρατσιστικές απόψεις υπάρχουν σίγουρα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί οι κυβερνήσεις να τις πυροδοτούν με τα χρήματα των φορολογωμένων. Οι κυβερνήσεις ε, ε, πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και πρέπει να το κάνουν αυτό. Αλλά η Ουγγρική κυβέρνηση δίνει ένα ανησυχητικό και πολύ επικίνδυνο παράδειγμα όσον αφορά τα θέματα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα μου δυστυχώς έχει γίνει παράδειγμα ανελεύθερου κράτους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε πώς ακολουθούν και άλλοι το παράδειγμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συγκεκριμένα στην Πολωνία, αλλά όχι μόνο εκεί. Ε, στη διάρκεια των ετών και φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες επί για πολύ σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, θέματα κράτους δικαίου στην Ουγγαρία, αλλά αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να ε, διορθώσουν τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Δεν μπόρεσα να αναφερθώ σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά ε, είναι καταγεγραμμένα. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στα εργαλεία που υπάρχουν για να διορθωθεί η κατάσταση, προτού να είναι πολύ αργά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Γκάμπερ από το Πανεπιστήμιο Πέξεν για την παρακολούθηση των μέσων μαζική ενημέρωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Με καλέσατε για να σας μιλήσω για την κατάσταση των ΜΜΕ στην ε, Ουγγαρία, των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ έχω διαφορετική γνώμη για την κατάσταση, ε, την ποιότητα της κατάστασης ε, με τον Ουγγρικό λαό από ό,τι ακούσατε μέχρι στιγμής από τον Υπουργό θα σας παρουσιάσω όμως και τα δικά μου επιχειρήματα. Πολύ συχνά με ρωτά αν υπάρχει ελευθεροτυπία σήμερα στην Ουγγαρία. Η απάντησή μου είναι ότι έχω, έχει μείνει κάποιο ελεύθερο τύπο, αλλά δεν έχουμε ελευθεροτυπία. Γιατί η ελευθεροτυπία σημαίνει πολύ περισσότερο από τον αγώνα κάποιων ε, ελάχιστων ε, ε, θαραλέων δημοσιογράφων. Ελευθερωτική είναι μια κατάσταση όπου όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν ίσες ευκαιρίες ε, να εκφραστούν και το ακροατήριο έχει ισότιμη πρόσβαση σε διαφοροποιημένη πληροφόρηση και το ΦΙΔΕΣ για να προσπαθεί να νομοποιήσει την πρακτική για τα μέσα μαζικής ενημέρωση, επιχειρηματολογώντα ότι θέλει να δημιουργήσει μια ισορροπία των ΜΜΕ. Με άλλα λόγια, θέλει υποτίθεται να ενισχύσει τη θέση των φιλοκυβερνητικών μέσων μαζική ενημέρωση έναντι της υποτιθέμενης ε, ε, δεσπόζουσα θέσης των αριστεριζόντων ή φιλοσοσιαλιστικών ε, ΜΜΕ. Έτσι όμως και υποτίθεται ότι έτσι θα δημιουργήσει νέες προπτικές και πιο πλούσια δημόσια συζήτηση. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, γιατί αυτή η ισορροπία των ΜΜΕ ουσιαστικά γίνεται μέσω περιορισμού της χρηματοδότησης σε συγκεκριμένα ΜΜΕ και επίσης περιορίζει τον ζωτικό χώρο συγκεκριμένων μέσω μαζικής ενημέρωση. Αυτό είναι τα θεμέλια μιας πολιτικής ΜΜΕ, που θεωρεί τα ΜΜΕ ως μοναδικό μέσο πολιτικής επικοινωνίας. Και κάθε ε, η κρισή κριτική τη θεωρεί ως ε, επίθεση η κυβέρνηση. Προσπαθεί ε, να στιγματίσει τους επικριτές ε, χαρακτηρίζοντας τους προδότες ή ξένους πράκτορες όπως γνωρίζετε. Και πιστεύει σε αναφυσβήτητες βεβαιότητες η κυβέρνηση και όχι σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα. Το ουγγρικό σύστημα από το 2010 και μετά έχει υποστήριξει και έλευθε αλλαγέ. Η οικονομική κρίση του 2008 αποδυνάμωσε ιδιαίτερο στην αγορά διαφήμιση και ω εκ τούτου δεν είναι αρκετά προσοδοφόρο για του ε, δυτικού επενδυτέ. Ξένοι όμιλοι και εταιρείε που είχαν μετοχές ε, ε, στα μέσα μας και σε ενημέρωση τη Ουγγαρία, όπω η Deutsche Telekom ε, ήξερα ότι θα του παρακολουθούσαν οι επιχειρηματίε με στενού δεσμού με το κόμμα Φίδε. Ο Άντρι Βάινερ τη ε, Μια Κυβερνητική Επιτροπή, ε, είναι ε, ισχυρός ε, πολιτικός, επίσης Σάρος, ε, φίλος του Πρωθυπουργού και Άντα Μότουετζη, γιο του Προέδρου της ε, Ουγγρική Εθνική Τράπεζα. Θα σας παρουσιάσω μερικά πραγματικά περιστατικά για το σύστημα του μέσου μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία σήμερα είναι ψηφιδωτά ενός ευρύτερου ψηφιδωτού που χαρακτηρίζει, χαρακτηρίζεται από μια ήπια λογοκρισία. Ε, είναι μια προσπάθεια του ΦΙΝΤΕΣ να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τις ψηφιακές πλατφόρμες, στους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, μέχρι και τη διανομή των εφημερίδων ε, βέβαια αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, στα ΜΜΕ προέρχονται από συστηματικές πολιτικές παρεμβάσεις. Πρώτο παράδειγμα, μία, ένα από τα βασικά ε, ε, δυτικά κανάλια ανήκουν στον Άντριο Βάινορ. Επίσης είναι ε, ο ιδιοκτήτης του μοναδικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που έχει και τοπικές ε, και εθνικές ε, εφημερίδες και έχει σκανδαλοθυρικό τύπο. Μέχρι το 2014 δεν είχε καμία παρουσία στην αγορά ΜΜΕ. Η TV2 είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος αποδέκτης κρατικών διαφημίσεων και η επιτυχία του στον κλάδο αυτό είναι δυσανάλογη με το μερίδιο αγοράς. Σε σχέση με το RTL, RTL Club που είναι ο βασικός ανταγωνιστής, ε, το κράτος ε, ε, ξοδεύει κοσαπλάσια κονδύλια για να διαφημίσει στο κανάλι του Σάμορ, το TV2. Επίσης, ο Χάρη Πέτσενερ έκλεισε την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Εθνική Εφημερίδα που ήταν επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση και ε, μάλιστα υπέστηκε πολλές έρευνες. Έκλεισε χωρίς καν προειδοποίηση αυτή η εφημερίδα. Δύο εβδομάδες μετά ε, ο ιδιοκτήτης 12 ε, περιφερειακών ε, περιφερειών, περιφερειακών εφημερίδων που πουλήθηκε σε ένα φίλο του Πρωθυπουργού. Και ο Μέιν Σάρος έγινε ιδιοκτήτης ξαφνικά 12 περιφερειακών εφημερίδων, περιοδικών, τηλεοπτικών σταθμών και μερικών τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, ε, μόνο το 2016 είχε 340 εκατομμύρια τζίρο, ενώ πριν το 2014 ήταν ανύπαρκτος στην αγορά με μία εψίλον της, της Επίση, Επίσης, μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα λαμβάνει περίπου το 90% των εσόδων από κρατική διαφήμιση, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για το πόσο βιώσιμη είναι η εφημερίδα αυτή. Το ίδιο ισχύει και για κάποια περιοδικά. Ε, ένα περιοδικό που ελέγχει ο Μέισαρος ε, αντλεί τα μισά έσοδα από κρατικές διαφημίσεις. Η διανομή τέτοιων κρατικών διαφημίσεων δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος ή τη, τη σύνθεση του ακροατηρίου. Και ουσιαστικά είναι παράνομη μορφή κρατικής ενίσχυσης. Μάλιστα το ενωσιακό δίκαιο προβλέπει τέτοια μέσα για να αποκατασταθεί μια στρεβλωτική για την αγορά κρατική ενίσχυση που παραβιάζει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που έγινε στις αρχές του 2017 προέκυψε ότι τα ΜΜΕ που συνδέονται με το κυβερνητικό κόμμα προωθούν τις κυβερνητικές πολιτικές και είναι πολιτικά όπλα κατά ιδιωτών, κομμάτων ή ομάδων που δεν είναι της ε, κυβερνητικής αρεσκίας. Επίσης, οι οργανώσεις φιλοκυβερνητικών μέσω μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα συντονισμό μεταξύ τους και ανταλλάσσουν και πληροφορίες. Η μεταρρύθμιση της αγοράς ΜΜΕ στην Ουγγαρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις μεροληπτικές αποφάσεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που συστήθηκε με έναν επίμαχο νόμο του 2010 και που απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη που έχουν διοριστεί από το κόμμα Φίδες και οι αποφάσεις αφορούν την κατανομή του ραδιοφάσματος και την έγκριση συγχωνεύσεως στην αγορά ΜΜΕ. Ε, επίσης, ε, έχει διασυνδέσεις ε, με επιχειρηματίες ε, του κυβερνώντος κόμματος. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα έχουν την ευκαιρία να ορίσουν την ανεξαρτησία όχι ως προαπαιτούμενο. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δίνονται τα μέσα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποφάσεων και των ενεργειών των αριθμιστικών αρχών. Τα μέσα ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής, στα μέσα, στα, στην οδηγία μέσων, τα κρατικά μέσα θεωρούνται ως εγγυητές της πολυμορφίας, αλλά πολύ εύκολο είναι να μετατραπούν στους ε, ε υπηρέτες των κυβερνητικών αναγκών. Επίσης, η εντολή της δημόσιας υπηρεσίας δεν είναι διαφανής, ούτε υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Γι' αυτό και μπορεί να γίνει υποχείριο ε, πολιτικών ε, παιχνιδιών. Επίσης, παραβιάζεται και η οι ενωσιακές ενισχύσεις για τις κρατικές ε, οι, οι ενωσιακοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις γιατί σίγουρα οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται από το κυβερνό κόμμα δεν ε, σέβονται αυτούς τους κανόνες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αποφασιστικά να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής ένας από του σημαντικότερου, ενός από τους σημαντικότερους φορείς της κρατικής προπαγάνδας στην Ουγγαρία. Ε, είχαμε κάτι αντίστοιχο και στην Ιταλία. Ε, με μονοπόλιο των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που ουσιαστικά ξεριζώνουν κάθε μορφή αυτονομίας. Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την κατάσταση στα ουγγρικά ΜΜΕ που κρατά χρόνια τώρα δείχνει πως μια αυταρχική κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσκήνιο. Βέβαια, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ε, μόνο απλά λόγια. Θέλουμε μια ξεκάθαρη δράση. Ευχαριστώ. Thank you. And now we give the floor to the final speaker. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μίκλος Σάντο από το Κέντρο Θεμελιδών Δικαιωμάτων Διευθυντής. Παρακαλώ και εσείς 10 με 12 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω, για την πρόσκληση. Είμαι διευθυντής ενός κέντρου δημόσιων αναλύσεων και μελετών. Και υπό αυτήν την ιδιότητα θα σας μιλήσω για πολιτικά για τα πολιτικά δρόμενα και την πολιτική κατάσταση στην Ουγγαρία ίσως φωτίσω διαφορετικά κάποιες πτυχές. Πάντως όπως και αν έχει. Χαίρομαι ιδιαίτερως που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρότεινα να πάμε πίσω στην αρχή, στο 2010 και στις γενικές εκλογές που έγιναν εκείνη τη χρονιά. Ίσχυε τότε ο προηγούμενος εκλογικό νόμος, είναι παρόμοιος με τον ε, νυν ισχύοντα, ένα μεικτό σύστημα προς ε, προβλέπεται πήραν την πλειοψηφία των δύο τρίτων ε, τα δύο κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, ο κόσμος ήξερε τι ψήφιζε. Δηλαδή, ότι αν ψηφίσει κάποια μεμονωμένα άτομα, δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία ο Βίκτορ Όρμπαν, αλλά πλειοψηφία των δύο τρίτων. Το γκρικό σύνταγμα και οι συνταγματικέ παραδόσει. προβλέπουν ότι με την πλειοψηφία των δύο τρίτων είναι, υπάρχει δυνατότητα τροποποίηση του συντάγματο και τη θεμελιώδη νομοθεσία. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί τα περισσότερα από τα ζητήματα που έχουν αναφερθεί σήμερα στη συζήτηση έχουν να κάνουν με μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2010 ή το 2011. Το νέο κοινοβούλιο πράγματι τροποποίησε το Σύνταγμα, τέλο πάντων ενέκρινε νέο Σύνταγμα, ενέκρινε νέο νόμο για τα μίντια, μεταρρύθμισε τον εκλογικό νόμο και πολλούς νόμους που αφορούσαν τη λειτουργία ε, του δικαστικού συστήματος. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολλή ώρα. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, έγιναν αντικείμενο δρυμίας κριτικής και σε εσωτερικό επίπεδο και ιδίω από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης βέβαια και τους διανοουμένους από όλες τις πλευρές πολιτικού αλλά και στο εξωτερικό. θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει οφθαλμαπάτη το ότι μπήκε στο προβολέα της δημοσιότητας η Ουγγαρία με όλες αυτές τις διαδικασίες ε, παραβιάσεων. Κοίταξα εγώ τις ε, στατιστικές για τα τελευταία δέκα χρόνια και τις διαδικασίες ε, παραβάση. Η Ουγγαρία ούτε στην πρώτη, ε, ούτε στην κορυφή, ούτε στη βάση της πυραμίδας είναι σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες, σε που έχουν κινηθεί. Και με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα πιο πρόσφατα του 2016, 1570 είναι οι διαδικασία παραβάση 57 αφορούν την Ουγγαρία, άρα στη 16, η θέση είμαστε. 6,3% δηλαδή των υποθέσεων αφορούν τη χώρα μας. Βέβαια, υπάρχουν δυναμικές διαμάχες ε, και αντιπαράθεση μεταξύ του εθνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αλλά δεν είναι κάτι πολύ πιο περίεργο και οξυμένο σε σχέση με το τι μπορεί να συμβαίνει με την Γερμανία ή άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η βάση αυτή τη συζήτηση. Οι πολιτικέ αυτέ διαδικασίε και οι κριτικέ κατά τη Ουγγαρία και οι διαδικασίε παραβάσει που έχουν κινηθεί κατά τη Ουγγαρία βασίζονται στο εξή. Και αυτό είναι και το θεμελιώδε ζήτημα. Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και η Ουγγρική Κυβέρνηση έλαβαν τι αποφάσει αυτέ το θέμα είναι, είχαν το δικαίωμα να τι λάβουν, ναι ή όχι αυτέ τι αποφάσει. Γιατί μια πλευρά λέει ότι πρόκειται για ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Άρα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν και την αρμοδιότητα να παρακολουθούν και να επιβλέπουν αυτές τις αποφάσεις. Αυτό όμω δεν είναι συζήτηση για το κράτο δικαίου και τη δημοκρατία, αλλά μια συζήτηση για την εθνική κυριαρχία. Δυστυχώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι σαφές ούτε από πολιτικής και νομική πλευράς τι συνιστά αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα και τι συνιστά ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για πολλά μείζωνα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. ζητούνται τα θέματα όχι μόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε κάποια συνταγματικά δικαστήρια για ε, το, τη συμβατότητα ε, των ε, εθνικών νομοθεσιών με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι αρχές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά υπάρχουν και κάποια συνταγματικά δικαστήρια σε κράτη-μέλη της Ένωσης που έχουν άλλη άποψη, ότι και αυτά δηλαδή μπορούν να αποφανθούν. Γιατί ξέχασε. Γιατί λησμόνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Αρχικά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προηγούμενα σχήματα ξεκίνησαν ως ε, ένας χώρος οικονομικής συνεργασίας σε περίοδο οικονομικής άνθησης και τα πιο πολλά ζητήματα αφορούσαν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, εμπνευμάτων κτλ. Υπήρξε αναρμόνιση πολλών κανόνων που πλέον αποτελούν τμήμα της δευτερογενούς νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. επαναλαμβάνω, σε συνθήκε οικονομική άνθηση. Εκεί ξεκίνησαν αυτά τα ζητήματα και αποχώρησε τη Δυτική Ευρώπη. Οπότε τότε ποτέ δεν είχε ανακύψει θέμα εθνική κυριαρχία. Δεν συζητούνταν τέτοια θέματα. Όμως τα τελευταία 10-15 χρόνια και παραπάνω όλο και περισσότερε προκλήσει αναφύονται που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχώρησαν οι πρώην χώρες, εντελώς διαφορετική η νομική και πολιτιστική του κουλτούρα και τέλος διαφορετική αντίληψή τους για την εθνική κυριαρχία. Σκεφτείτε το. Μια χώρα που πανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1989 είναι προφανές ότι οι εθνικέ αρμοδιότητε, η εθνική κυριαρχία, ο όρο έθνο σημαίνει κάτι εντελώ διαφορετικό από μια χώρα που ποτέ δεν βίωσε ένα κομμουνιστικό καθεστώ για μισό αιώνα. Φυσικά υπήρξαν οικονομικέ και πολιτικέ κρίσει ο πολιτικός ρόλος, αρήτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συρρυκνώθηκε. Η όλη ευρωπαϊκή συνταγματική διαδικασία είναι ένα θέμα επίσης και βέβαια και η καυτή πατάτα. Τα ζητήματα της μετανάστευσης ε, και της λαθρομετανάστευσης ε, έχουν πλέον περιπλακεί πολύ περισσότερο και αποτελούν πρόβλημα σε μια εποχή που δεν έχουμε πλέον την οικονομική άνθηση και ευημερία του παρελθόντος. Και τώρα λοιπόν ανακύπτουν και οι συζητήσεις για την εθνική κυριαρχία και τις εθνικές αρμοδιότητες. Η συζήτηση αυτή γίνεται τώρα λόγω ακριβώς όλων αυτών των προκλήσεων. Και έχει μπει στο προσκήνιο αυτή η συζήτηση. λύσει που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιε φορές δεν ικανοποιούν. Γι' αυτό και κάποια κράτη-μέλη θεώρησαν ότι και τα ευρωπαϊκά αλλά και βέβαια κυρίως τα εθνικά προβλήματα μπορούν να τα επιλύσουν με εθνικέ πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Οι οποίε λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και έχουν να κάνουν κυρίως με τη δημόσια πολιτική. Επηρεάζουν το σύνολο τη κοινωνία αυτέ οι αποφάσει. Μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, έχουν τέτοιου είδους αρμοδιότητες ή όχι και πρόκειται μόνο για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Όταν μιλάμε για εθνική κυριαρχία, πρέπει να δώσουμε απάντηση στο εξή ερώτημα. Πίσω από όλες αυτές τις διαφορές για το πώς κανείς αντιλαμβάνεται την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, υπάρχουν και ζητήματα κοσμοθεώρησης, πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Τον Ιανουάριο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέδωσε μια γνωμοδότηση. όπου αναφέρεται ότι οι ιδρυτικές συνθήκες ε, δεν παρέχουν ένα σαφή ορισμό για τις θεμελιώδεις αρχές σε ό,τι αφορά τα όρια της εθνικής αρμοδιότητας και το κατά πόσο θα πρέπει οι ευρωπαϊκές αξίες να σέβονται την εθνική ταυτότητα και τούμπαλιν η εθνική ταυτότητα, ευρωπαϊκές αξίες, πολλές φορές ε, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο. Κάποιοι λένε ότι χρειαζόμαστε μία ε, πλουραλιστική Ευρώπη με ισότητα, διαφορετικότητα. Άλλοι λένε ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα σέβεται την εθνική κυριαρχία και τις εθνικές αρμοδιότητες. Το πρόβλημα είναι ακριβώς να επιλύσουμε τη σύγκρουση αυτή μεταξύ αυτών των δύο. Την Ευρώπη των εθνών ή τα κράτη-έθνη. Τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο Λούτσακ για, για το κράτος δικαίου. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσουμε για πολλά και να συζητήσουμε για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Έτσι θα ήμασταν πιο ειλικρινεί μεταξύ μα και θα λύναμε προβλήματα. Σε μια τέτοια συζήτηση ευχαρίστω να συμμετέχω. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στα μέλη και θα ξεκινήσω με του ε, συντονιστέ. Σα παρακαλώ απλώ ε, Ε, να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ε, σκιώδεις ηγητές οι οποίοι αντικαθίσταται από μέλη. Αυτά όλα είναι προαποφασισμένοι. Ε, πολύ αυστηρό χρονικό όριο, δύο λεπτά ο καθένας. Ε, θα σας κόψουμε στο τέλος του καταλόγου, αν βρίσκεστε στο τέλος του καταλόγου, γιατί πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τις 11 παρα 20. Μην απογοητευτείτε αν δεν μπορέσετε να μιλήσετε, θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τους πάντες. Πολύ αυστηρά λοιπόν, δύο λεπτά, το έλκ και η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που εκπροσωπείτε στην Επιτροπή μας εδώ, την Ουγγρική Κυβέρνηση. Και πάντοτε, ακόμη και όταν είναι δύσκολα τα ζητήματα, έρχεστε εδώ για να ακούσετε ερωτήσεις και να δώσετε απαντήσεις. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μην θέλουν να έρθουν ή όπως και στην Επιτροπή ε, για τον Παναμά, για τα έγγραφα Παναμά, ε, ναι μεν ήρθαν αλλά δεν έδωσαν απαντήσεις. Επίσης σέβομαι ε, αυτό που είπατε για τις διαδικασίες ε, παραβίασης ε, των συνθήκων. Υπάρχει μια αντίθεση εδώ σε σχέση με την πολωνική κυβέρνηση που έχει υποδεχθεί την Επιτροπή της Βενετίας Υπάρχει ένα πρόβλημα ε, γιατί εσείς έχετε δώσει ένα καλύτερο παράδειγμα. Μπορεί να ε, μην συμφωνώ μαζί σας εγώ, αλλά γιατί εσείς δέχεστε αυτό που κάνει η Πολωνία και το υποστηρίζετε. Γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί σε ό,τι αφορά την Επιτροπή της Βενετίας και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό το οποίο επίσης σέβομαι και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό είναι η οικονομική ανάπτυξη που πλέον ε, φτάνει και σε ένα στρώμα του πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν είχε επωφεληθεί. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα στατιστικά στοιχεία και από τα νούμερα σε ό,τι αφορά τους μισθούς, ιδίως ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν ε, ανεβεί 14% τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Και έχουμε και θετικές κοινωνικές εξελίξεις εκ νέου. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί και οι αλλά και άλλοι οργανισμοί που μετρούν αυτά τα σχετικά έχουν ε, δώσει θετική αξιολόγηση. Όμως, εκεί που βλέπω εγώ πρόβλημα είναι αυτή η αδιάκριτη μεταχείριση της νόμις μετανάστευσης και από την άλλη της ε, μετανάστευσης και τις σχέσεις με την τρομοκρατία για παράδειγμα. Και τα λέω πολύ ξεκάθαρα. Οι τρομοκράτες πράγματι χρησιμοποιούν όλες τις διόδους ε, και μέσω της ε, παράνομης μετανάστευσης αλλά και μέσω της νόμιμης οδού με αεροπλάνα, πλοία, σιδηρόδρομο έχουν κοινωνικές διασυνδέσεις δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια, στο ίδιο καλάθι ε, τους μετανάστες με τους τρομοκράτες ε, και είναι πραγματικά παράδεκτο να θεωρείται αυτομάτως ο μετανάστης ε, και τρομοκράτης και πρέπει το αφήγημα αυτό να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αυτό το αφήγημα πλέον στην Ουγγαρία. Ναι, έπρεπε να είμαστε αυστηροί στα δύο λεπτά. Είχα να πω και κάτι ακόμα, αλλά πρέπει να είστε όλοι πάρα πολύ πειθαρχημένοι, λέει ο πρόεδρο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Ο κύριο Νόιντρου για το σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Μία, ε, κύριε Υπουργέ, κάποιες σύντομες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Στις 27 Οκτωβρίου στο κρατικό ραδιόφωνο ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι όλες οι οργανώσεις ε, οι οποίες αποκαλούνται οργανώσεις Σόρος θα πρέπει να παρακολουθούνται από τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση ε, παρακολουθεί ε, τις επιχειρήσεις αυτές ε, οι οποίες θεωρείται ότι σχετίζονται με τον κύριο Σόρο. Ε, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι η αντιπολίτευση είναι τμήμα των δημοκρατικών θεσμών, αλλά είναι ξένοι πράκτορες, εχθρός, οι οποίοι απειλούν ε, ε, την εθνική ασφάλεια. Δεύτερη ερώτηση. Ε, κάποιος πριν με λίγες ημέρες εδώ στις Βρυξέλλες είπε ότι αυτές οι ακροάσεις ε, στην πραγματικότητα είναι κυνήγι μαγισσών και ότι του υπενθυμίζουν τις ε, ψευδοδίκες ε, του κομμουνισμού. Πιστεύετε ότι πρόκειται για κυνήγι μαγισσών εδώ, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια ψεύτικη δίκη του κομμουνισμού. Ευχαριστώ. Για την ομάδα του ECR, η κυρία Στίβενς, παρακαλώ. Η κυρία Στίβενς, ε, ο κύριος Γιούρεκ εκπροσωπεί την κυρία Στίβενς. Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Και σίγουρα το ότι ακούσαμε διχασμένες γνώσεις είναι περίτρανη απόδειξη της πολυμορφίας, της πολυφωνίας και του πλουραλισμού. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό να μας παρουσιάσει ε, για τα οικονομικά αποτελέσματα μας μιλήσατε για κάποιες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών, των μίντια και ε, μερικές φορές ε, παρασυρώμαστε από την ε, θέση και τις επικρίσεις αντιπολίτευσης, αλλά συχνά δεν ακούμε παρκώς τις απόψεις της κυβέρνησης. Πείτε μας λοιπόν γιατί ακριβώς έγιναν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή της ε, ε, του Ελσίνκη. Μιλήσατε για έλλειψη στην ελευθερία των δραστηριοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τη δική σα επιτροπή του Ελσίνκη. Μπορείτε να το τεκμηριώσετε. Και επίση τον καθηγητή, θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Πόλιακ και να μου πει πώ λειτουργούσε η πολιτική διαφήμιση ε, κατά τη διάρκεια των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων τότε υπήρχε ισότιμη διαφήμιση σε όλες τις εφημερίδες άσχετα με την πολιτική απόχρωση, την πολιτική παράταση. Και τώρα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Και προς τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Σάντο, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, οι ΜΚΟ στην Ουγγαρία έχουν διαφοροποιημένη θέση. Μπορούμε να πούμε ότι όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Ουγγαρία είναι ε, επικριτικές κατά της κυβέρνησης. Ή υπάρχουν και κάποιες που δεν συμμερίζονται τις δικές απόψεις. Επίσης, ε, κυρία Χολμάιερ, στη πατρίδα σας, στη Βαβαρία, η δράση της κυβέρνησής γιατί προσέξτε όταν μιλάτε για την Πολωνία, θα σας διακόψω γιατί ε, κανείς δεν θα επερβεί τα δύο λεπτά. Κανείς. Θέσετε τις ερωτήσεις σας, διακόπτω. Η σκιώδης των φιλελευθέρων, η ο κύριος Μισελ είναι ε, εδώ για δύο λεπτά. Εδώ και επτά χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία διαπράττει η κυβέρνησή σας που από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσβάλλουν τις συνθήκες και τις συνθήκες προσχώρησης τις οποίες εξ όσων γνωρίζω υπογράψατε ελεύθερα. οι ανταλλαγές που είχατε με τις ευρωπαϊκές αρχές και τα θεσμικά όργανα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά που κάνατε είναι ψευδή και προσβλητικά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Υπουργέ, ε, χρησιμοποίησατε το ίδιο ύφος ε, το προκλητικό και εδώ σήμερα. Ε, αναφέρεστε στη συμπεριφορά αυτή ενώπιον των πολιτών σας είναι άδικη συμπεριφορά και ορισμένες φορές σιωπείτε και δεν λέτε για παράδειγμα ότι η Ουγγαρία ε, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια που βελτιώνουν τη ζωή κάθε Ούγγρου και οι λεγόμενες εθνικές διαβουλεύσεις τις οποίες οργανώνουν οι αρχές σας όπως για παράδειγμα το Let's Stop Brussels ε, είναι μαρτυρία της χειραγώγησης και της ε, υποτίθεται δημόσια διαβόλευση για να υπερασπίσετε τις προθέσεις τη. Σήμερα λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι η αντίληψη που έχετε εσείς για τη δημοκρατία δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ευρωπαϊκές αξίες πλέον, ούτε στα κείμενα τα οποία ε, τις ε, ε, προσπογράφουν και πραγματικά διαπιστώνω ότι η αντίληψη που έχετε για τη δημοκρατία και τις ανθρώπινες αξίες οδηγούν χωρίς ε, καμία διαφορά σε μια συμπεριφορά μιας κυβέρνησης την οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ε, τυραννία κατά της πλειοψηφίας. Το άρθρο 7 ε, αναφέρεστε στον πραγματικό ειλικρινή διάλογο για να επιτρέψει να εγκρίνετε εσείς τις πολιτικές σας ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία δεχτήκατε όταν ε, προσχωρήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, σας καλώ να δεχτείτε αυτή τη διαδικασία που θα σας επιτρέψει να ε, με τιμή στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ, είναι απλή. Κάθε φορά λέτε ότι είστε διατεθειμένοι να συμμετέχετε στο διάλογο με τους Ευρωπαίους τους και ε, ε, ότι είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε το άρθρο 7.1. Για την ΚΟΕ, η κυρία βερσιά Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το δημοψήφισμα για να διαβουλευτούμε με του πολίτες μπορεί να είναι καλό. Και λυπάμαι στη Γαλλία, δεν λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2005 και λυπάμαι γι' αυτό ω Γαλλίδα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνεται συζήτηση και όχι να χειραγωγείται το, η κοινή γνώμη. Ε, θα πρέπει να ε, έχουμε ερωτήσεις ε, οι οποίες πρέπει να μας απαντώνται όταν πρόκειται για λεπτά θέματα όπως αυτό τη μετανάστευση και συμφωνώ με αυτό που είπε και η κυρία Χολμάγερ σε αυτό. Θα ήθελα να σας θέσω την εξής ερώτηση. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι ε, υπάρχουν ε, αρκετοί ετούνται σε στην ε, ε, Ουγγαρία και το πολύ μικρό αριθμό αιτήσεων που γίνεται αποδεκτές, που είναι από τους μικρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς δικαιολογείται τις επιθέσεις κατά των κυβερνητικών οργανώσεων που φροντίζουν αυτούς τους πρόσφυγες στην Ουγγαρία και κυρίως στα σύνορα οι εκστρατείε που συνοδεύουν τι διαβουλεύσεις είναι πάρα πολύ επιθετικέ κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονό ότι είστε ε, από τους ανθρώπους που, από τις χώρες που χρηματοδοτούνται καθαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σχέση 1 προς 5. Πώς ε, θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε έναντι των υπολείπων Ευρωπαίων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι καθαροί φορής προ την Ουγγαρία. Τι σημαίνει για σας η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας. Πώς ενθαρρύνετε εσείς τη δημοκρατία στις οργανώσεις τη κοινωνίες, των πολιτών, στη κοινό βίο ε, και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Οι καλές και οι κακές σχέσεις ε, φαίνεται να είναι ουσιαστικά το νήμα το οποίο κινεί την ε, Ουγγρική κυβέρνηση και θα ήθελα να ρωτήσω και τις οργανώσεις τι συγκεκριμένες δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Τέλο, όταν η Ουγγαρία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσχώρησε και στι αξίε, της. καθολικέ αξίε, όπω καθορίζονται από το άρθρο 2, είναι τα κριτήρια τη Κοπενχάγης, τα οποία βασίζονται σε διεθνεί συμβάσει και πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και υπάρχουν κανόνε κανόνες και ε, αυτά όταν τα αμφισβητείτε δεν αμφισβητείτε και τη συμμετοχή σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρου των Πρασίνων, το λόγο κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στην κυρία Παρδάβη από την Ουγγρική Επιτροπή του Ελσίνκη. Ποια είναι τα αποτελέσματα της νομοθεσίας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα προβλήματα με την ξένη χρηματοδότηση και το πώς επηρεάζει τους Ούγγρους πολίτες ε, που βοηθάτε μέσα στη χώρα. Πώς σας επηρεάζει λοιπόν αυτή η νομοθεσία για τις ΜΚΟ. Δεύτερη ερώτηση προς τον, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Έχουμε την υπόθεση Μπάκα κατά της Ουγγαρίας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, η απόφαση του δικαστηρίου έλεγε αποκατάσταση των δικαστών και επαναφορά τους στο δικαστικό θόκο στα ουγγρικά δικαστήρια εφαρμόστηκε η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ουγγρική κυβέρνηση. Τι συνέχεια δόθηκε. Ερώτηση προς τον κύριο Σάντο. Με προβλημάτισαν τα λεγόμενά σας. Λέτε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες που περιχαρακώνονται στο άρθρο 2 αλλά να διατρέξουν τον κίνδυνο να υποστούν τις κυρώσεις στο άρθρο 7. Θεωρείτε ότι είναι σχετικές οι ευρωπαϊκές αξίες και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τα ήθη και έθιμά τους. Ή λέτε ότι το άρθρο 2 της Ηθίκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άρθρο που θα πρέπει να εφαρμόζουμε και να σεβόμαστε όλοι. Και η τελευταία ερώτηση πάλι προς τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, γιατί η Ουγγαρία ε, ζήτησε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, κόπτεστε τόσο πολύ για την ε, εθνική κυριαρχία, αν τη θεωρείτε τόσο σημαντικό. Και γιατί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει κάποια διαφοροποίηση της κυριαρχίας, ιδιαίτερα για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουίμπερκ από τον EFTD. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό που είχε την καλοσύνη και ήρθε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση και η Ουγγρική κυβέρνηση ε, έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί πολύ αποτελεσματικά στις ε, επιταγές των Βρυξελών και τη συγχαίρω για την αντίστασή της. Ιδιαίτερα αντιστέκεται στη, στο μεταναστευτικό δίκαιο που προσπαθεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά είστε παράδειγμα προς μίμηση και για μας. Γιατί δεν ασπάζεστε το μοντέλο της ε, πολιτιστικής πολυμορφίας αλλά εκπροσωπείτε και προσπίζετε τη θέση ε, του Ουγγρικού λαού, των συμπολιτών σας. Μακάρι να είχαμε Υπουργό Μετανάστευσης σαν και εσάς και στην πατρίδα μου τη Σουηδία. Και αυτά που ακούμε για το τι συμβαίνουν στα άλλα κράτη-μέλη δεν είναι εφαλκιδευμένες ειδήσει, δεν είναι fake news. Δείτε την κατάσταση στη Σουηδία σήμερα. Βλέπετε πώς ξένους μαχητές ε, έχουμε. Έχουμε συνοικίες που η κατάσταση ασφάλειας είναι πολύ ανησυχητική αν θέλουμε να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα του πολίτη να νιώθει ασφαλής όπου και αν βρίσκεται. Και αυτό το δικαίωμα έχει υπονομευθεί. Κύριε Υπουργέ, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζέλστρα που μου παραχώρησε το χρόνο αγόρευση του, να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του και να σα ευχαριστήσω που ήρθατε για μια ακόμη φορά για να απαντήσετε σε τελείω ανεδαφικέ, ανυπόστατε και παράλογε κατηγορήσει βάρο τη κυβέρνησή σα. Εσεί προσπαθείτε να προσπίσετε την, την εθνική ταυτότητα και την ασφάλεια των Ούγγρων και αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Και ε, είστε κατά των επιταγών των Βρυξελών για τη μετανάστευση, χωρίς καμία παραβίαση των συνθήκων. Και οι κατηγορίες για αντισημιτισμό είναι παράλογες. Ο ίδιος ο Νετανιάχου τις κατέριψε αυτές τις κατηγορίες ε, και η Ισραηλινή κυβέρνηση πρόσφατα υπενθύμησε ότι η, η επίκριση κατά του κυρίου Σόρου είναι απόλυτα νομότυπη, γιατί ο κύριος Σόρου συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση ε, και διεκδικεί το 1 εκατομμύριο παράνομο μεταναστών και την ε, είσοδό του, νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατία και πολύ σωστά μα τα είπατε. Το επισήμανε και στον κύριο Φερχόφστατ στη συζήτηση τη διάσκεψη των Προέδρων. Και ταυτόχρονα η απέτηση διαφάνεια για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ είναι απόλυτα θεμητή. Πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, ιδιαίτερε χώρε του Νόσου, είναι συνένοχοι των λαθροδιακινητών και τη μαφία. Είναι σημαντικό να θέλετε να αποκαταστήσετε τη διαφάνεια στη λειτουργία του. Ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία, ο κύριος Πόλιακ, ε, ε, τι ελευθερωτική είχαμε στη Γαλλία όταν στις ε, προεδρικές εκλογέ όλα τα ΜΜΕ ήταν υπέρ του κύριου Μακρόν και κανένα δεν προωθούσε την κυρία Λεπέν. Επίση, είδαμε την προηγούμενη σοσιαλιστική ουγγρική κυβέρνηση και τι βίε καταστολές κάποιων διαμαρτυριών για την εξέγερση της Βουδαπέστης. Αυτά γιατί δεν τα καταδικάσατε η κυβέρνηση Ορμπάν, Φίδες και οι δημοκρατικές ε, βλέψεις ε, του γκρικού λαού δεν γίνονται δεκτές δυστυχώς. Συγχαρητήρια πάντως εσύ για, για την υπομονή σας και σας ε, θέρμο παρακαλώ να συνεχίσετε την οξυδερκή αυτή πολιτική και να συνεχίσετε την δράση σας υπέρ της αφύπνισης των ευρωπαϊκών λαών. Βάιτεν Χόλτζερ, παρακαλώ, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ δεν κάνουμε κανένα σοου. Ε, εδώ ε, έχουμε πράγματι ένα χώρο διαλόγου και χαίρομαι που το τονίσατε και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για μια δίκη κατά της Ουγγαρίας ε, ή οποιαδήποτε ε, καταγγελία απέναντι στη χώρα σας. Μιλάμε για τις κοινέ αξίες και πρέπει να εστιάσουμε στις διάφορες χώρες και όχι ίσως μόνο στην Ουγγαρία. Εγώ θέλω να πω το εξή. Πράγματι έχουμε το θέμα των προσφύγων. Πήγα στο Ρότσικε και είδα εκεί πώς λειτουργούν τα πράγματα και πρέπει να σας πω πραγματικά ότι έμεινα ε, πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Έχουμε συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν βλέπω δηλαδή να μπορεί να θεωρηθεί θέαμα αυτό να μεταφέρονται με χειροπέδες έγκυες γυναίκες στο γιατρό. Δεν, δεν, μπορώ αυτά τα πράγματα να τα φανταστώ. Ε, και από ό,τι φαίνεται... Ε, Ε, να ε, λειτουργεί αυτό το μέτρο για το σεναριακό έλεγχο όσων 10.000 άτομα έχουν περάσει ε, στην Ουγγαρία. Σε ό,τι αφορά τώρα το μηχανισμό μετεγκατάσταση, είπατε και πολύ σωστά ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, αλλά γιατί δεν την τηρείτε τελικά αυτή την απόφαση. Και γιατί στο Συμβούλιο όταν έχετε κάποιες επικριτικές απόψεις γιατί δεν αναφέρετε στο Συμβούλιο μία πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώθηκε ο γύρος ε, με τους συντονιστές και τους ε, σκιώδεις και θα ε, περάσουμε στους υπόλοιπους. Της κυρία Γκάλη, πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δύο φορές έχουμε συζητήσει ήδη φέτος αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές μελέτες ε, ή δείκτες ε, που να έχουν δικαιολογήσει το λόγο που γίνεται για συστηματικές παραβιάσεις. Έχουμε το πίνακα βαθμολογίας, το scoreboard 17. Η Ουγγαρία είναι σχεδόν στην κορυφή του καταλόγου. Για δείτε αυτό το scoreboard για judicial review, να δείτε τι κάνουμε. Και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες παραβάσεις πάλι δεν είμαστε πάνω, είμαστε στη μέση. Και δεν έχουν ε, ασχοληθεί της Κομισιόν που κινούν διαδικασίες σε παραβάση ε, κατά τις με άλλες χώρες ε, που κάνουν τα ίδια. Και όσο ό,τι αφορά την Όλαφ ε, δεν βλέπουμε να υπάρχει διάθεση να δουν άλλες χώρες και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα μίντια και άλλες μεταρρυθμίσεις μας δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ από άλλες χώρες. Ο νόμος για τα μίντια, για παράδειγμα, πήρε το πράσινο φως τελικά μετά από τροπολογίες. Δεκάδες, χιλιάδες μήκυο υπάρχουν στην Ουγγαρία και λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Μία χούφτα είναι που έχουν πρόβλημα και αν δεν είχαν να κρύψουν κάτι, γιατί να μην δηλώνουν να παίρνουν πάνω από 30.000 ευρώ από ε, ξένη πηγή. Κανείς δεν δέρνει τους διαδηλωτές στην Ουγγαρία, δεν συλλαμβάνονται μέλη της αντιπολίτευσης δεν έχει σκοτωθεί κάποιο δημοσιογράφος, αλλά στα άλλα κράτη που εσεί δεν βλέπετε να υπάρχουν συστηματικά προβλήματα, έχουμε τέτοιε περιπτώσεις. Άρα είναι τυπικό, χαρακτηριστικό παράδειγμα διπλών δύο μέτρων και δύο σταθμών, απλά γιατί δεν ε, συμφωνούμε με τα σχέδιά σας ε, για την καταπολέμηση της μετανάστευση. Μια ακόμη δημόσια ακρόαση που σίγουρα θα εκνευρίσει πολύ τον ουγγρικό λαό. Κυρία Ιντβέλτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι μια πραγματική συζήτηση αυτή, λυπούμε που το λέω, αλλά ακούμε την προπαγάνδα τη Ουγγρική κυβέρνηση εδώ. Αλλά α μην αυταπατώμεθα, λέει ο Υπουργό, ναι, ναι. Νομίζετε ότι είναι αστείο. Ε, εντάξει, μπορείτε να είστε σαρκαστικό. Αλλά σα ακούμε, κύριε Υπουργέ, και λέτε εμεί οι Ούγγροι. Για να δούμε λίγο τα στοιχεία. Ε, εξ ονόματο ποιου μιλάτε, εξ όλων των Ουγγρών, όλου του Ουγγρικού λαού. Τη πλειοψηφία του γκρικού λαού. Γιατί αν δω τα στοιχεία, αν δω τα νούμερα, δεν κερδίσατε την πλειοψηφία στι τελευταίε εκλογέ και ο κύριο Όρμπαν δεν κέρδισε το δημοψήφισμά του. Άρα εκ μέρου ποιον μιλάτε τελικά. Προσπαθείτε να περισπάσετε την προσοχή μα από το γεγονό ότι ο κύριος Όρμπαν δεν έχει τελικά την πλειοψηφία και λέτε ότι ένα έθνο έχει το δικαίωμα να έχει τις δικές του θέσει. Εγώ, ξέρετε, διαφωνώ, διότι έθνο ε, δεν σημαίνει ένα πρόσωπο. Ο κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα στη δική του θέση. Γι' αυτό και στη δημοκρατία υπάρχει ο πλουραλισμό. Αυτό είναι ακριβώ αυτό που προσπαθεί να σκοτώσει το Φίντε και ο κύριο Όρμπαν. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Αν συγκρίνουμε τον ένα νόμο με τον άλλο και τη μια χώρα με την άλλη, μπορεί τα πράγματα να φαίνονται καλά. Ξέρουμε όμω όλοι μα ότι για 8 χρόνια τώρα ο κύριο Όρμπαν καταπιέζει και καταστέλει τι επικριτικέ φωνέ και την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι ψεύδο δημοκρατία. Λέτε επίση ότι οικονομικά τα πάμε πολύ καλά. Τι θα κάνει η Ουγγρική οικονομία αν δεν είχε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και η κυρία Βερζιά. Άλλοι πολίτε πληρώνουν για την οικονομική σα ευημερία. Λέτε λοιπόν ότι τα πάτε πολύ καλά και δεν θέλετε την υποστήριξη. Μα να το δούμε. σω να δούμε και τι γίνεται με τη διαφθορά και πόσα χρήματα κλέβει από τι τσέπε των Ούγγρων πολιτών. Και τέλο, νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα τα πολιτικά κόμματα να σταματήσουν να προστατεύουν τα μέλη του που δεν έχουν δημοκρατική συμπεριφορά. Και αυτό εδώ έχει να κάνει με το ΕΛΚΑ. Υπάρχουν και άλλε περιπτώσει όμως που άλλες πολιτικές ομάδες επίσης συμμετέχουν. Όμως, μετά από 8 χρόνια άκαρ που διαλόγονται εισαγωγικών με τον κύριο Όρμπαν, που δεν ακούει ε, τις φωνές ε, της δημοκρατίας, καιρό είναι πλέον ε, να διώξει κλωτσιδών το ΕΛΚ το Φίντες από τους κόλπους του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να συνεχίσω σε αυτά που έλεγε η κυρία Ινετφέλτ. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι κάνουμε επίθεση κατά των Ούγγρων, αλλά κάθομαι και δίπλα στο συνάδελφο εδώ, με τον οποίο συνεργάζομαι με μεγάλη ευχαρίστηση και είναι Ούγγρος. Και νομίζω ότι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να φροντίσει να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχίες ε, ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και επομένω και των Ούγγρων πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να παρέμβω όσον αφορά την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και κυρίως των γυναικών ε, της Ουγγαρίας. Η έκθεση για την υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών που δημοσιεύθηκε την Τρίτη λέει ότι στην Ουγγαρία η Ουγγρική κυβέρνηση ε, κατήργηση την ε, ε, αποζημίωση για αντισύλληψη, διότι ε, σκοπός είναι να αποφύγουν μη επιθυμητή εγκυμοσύνη. Ε, και επομένως αυτό επηρεάζει τα δικαιώματα των δικαιωμάτων και σας υπενθυμίζω ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ουγγαρία. Επίσης να σας πω ότι η έκθεση υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες μετανάστες χωρίς χαρτιά εξαιρούνται από όλες τις παροχές υγείας, που σημαίνει ότι οι έγκυες γυναίκες μετανάστες δεν έχουν έχουν πρόσβαση ε, και έχουν πρόσβαση σε γιατρό μόνο όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της γένας. Αυτό είναι απάνθρωπο. Τι μπορείτε να κάνετε ώστε όλοι οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ούγγροι πολίτες να προστατεύονται και να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός προστασίας. Υπήρξε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα συζητηθεί ε, τον επόμενο Μάρτιο για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και ε, τον Οκτώβριο του 2016 ε, ψηφίσαμε για να έχουμε ένα μηχανισμό για το κράτος δικαίου και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πριν από το Σεπτέμβριο του 2017 να γνωμοδοτήσει. Είμαστε στο Δεκέμβριο του 2017. Πότε θα ε, υπάρξει αυτός ο μηχανισμός για την κατάσταση του δικαίου για να γίνεται πραγματική παρακολούθηση του τι ακριβώς γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Κατζίσκα. Κύριε Υπουργέ, πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, χρειάστηκε να κάνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις πατρίδες μας, την Πολωνία, εμείς και την Ουγγαρία εσείς. Να εξασφαλίσουμε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, της ελευθερής έκφρασης, ε, του εκλογικού νόμου. Εσείς βέβαια ε, ανατρέψετε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, είχατε νέο καθεστώς ιδιοκτησίας, ε, ουσιαστικά έχετε ένα μονοκομματικό καθεστώς. Και έχω την αισθησία ότι ήρθατε εδώ σαν να ήρθατε σε πόλεμο. Ε, ότι θέλετε να αγωνιστείτε προς υπεράσπιση του γκρικού λαού. Κανένας δεν επιτίθεται όμω τον γκρικό λαό. Ε, σε τι κατά τη γνώμη σας συνίσταται η επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ουγγρικό λαό. Γιατί έχω πολλούς φίλους στην Ουγγαρία που αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία, αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου με τον τρόπο που το προβλέπουν και το κατοχυρώνουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες ψευδοεπιστημονικές ε, απόψεις και παρατραβηγμένοι ορισμοί δεν πρόκειται να το αλλάξουν. Δεν σας επιτίθεται κανένας, γιατί αντιμετωπίζετε τις Βρυξέλλες σαν να είναι Μόσχα και δημιουργείται μια εικονική κατάσταση, μια πλασματική κατάσταση ε, επικαλούμενοι κάποιες περίεργες ε, ε, επιρροές ε, των Βρυξελών και μία απόπειρα των Βρυξελών ε, να στερήσουν την ελευθερία από τον ουγγρικό λαό. Είναι δυνατόν. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρη. Δύο λεπτά παρακαλώ και εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απευθυνθώ στον Υπουργό. Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά και δεν είναι πρώτη φορά και δεν τυχαίο ε, και το έχουμε συζητήσει εδώ και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σε αρκετές περιπτώσεις ε, ότι επιδεινώνεται η δέσμευση της ε, κυβέρνησης της Ουγγαρίας στην οποία συμμετέχετε κι εσείς ενώπιον των αρχών για τις οποίες δεσμευθήκατε κατά την προσχώρησή σας το 2004 δίνεται ρεσιτάλ της ατζέντα της Ουγγρικής κυβέρνησης και μάλιστα ε, το λέτε επανειλημμένο. λες και εκπροσωπείτε όλο τον Ουγγρικό λαό. Μιλάτε συνέχεια για τους Ούγγρους και για το λαό της Ουγγαρίας, ενώ ε, είναι προφανές ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εδράζονται σε πολυφωνική δημοκρατία, σε ανοιχτή κοινωνία και εκεί χωρίς καμία αμφιβολία υπάρχουν και Ούγγροι που υπερψηφίζουν το Φιδές αλλά υπάρχουν και Ούγγροι που δεν ψηφίζουν υπέρ του Φιδές και εκπροσωπείται και αυτούς και αυτούς τους εκπροσωπεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι εξωτερική παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική στην οποία αναφερθήκατε. Είναι διάσταση των πολιτών των ε, εκατομμυρίων Ούγγρων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς δεν βρίσκεστε ενώπιον του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, βρίσκεστε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντάτε όσον αφορά τη δέσμευσή σα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει τη οποία κυρώσατε και την προσχώρησή σα το 2004. Και στην ευρωπαϊκή δέσμευση έχουμε κάθε δικαίωμα να ε, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου όταν βλέπουμε να ε, υποχωρεί η ελευθερία ε, της ενημέρωσης με συγκεκριμένη ε, απόφαση ε, νόμου. Όταν βλέπουμε να καταπιέζεται τα μέσα ενημέρωση τη Ουγγαρία, βλέπουμε την καταπίεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κυρίω όταν βλέπουμε ότι εσεί ε, θεωρείτε ότι υπάρχει απειλή κατά τη κυριαρχία τη Ουγγαρία, διότι η Ουγγαρία δεν τηρεί μια πολιτική μετανάστευση που είναι ευρωπαϊκή. Και αυτό έχει ε, ουσιαστικά καταργήσει την πολιτική ε, στην οποία συμμετέχετε. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλέσω τους υπουργούς και τους εκπροσώπους της Ουγγαρίας να μην θεωρούν ότι όλοι οι επικριτές ε, είναι πληρωμένα οι άνθρωποι του Σόρος. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλές επικρίσεις ε, ε, για τις προτάσεις του Σόρος, κυρίως όσον αφορά τον επαναπατρισμό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι, όσον αφορά τη διαβούλευση με τον λαό για το θέμα της μετανάστευσης, είναι ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι εάν ε, οι ερωτήσεις είναι παραπλανητικές, ε, τότε και η συνένεση ε, που θα λάβετε θα είναι παραπλανητική. Και αυτό φυσικά κάνει αυτό το ερωτηματολόγιο επικίνδυνο. Είναι παραπληροφόρηση όταν ο Ορμπάν λέει όταν σας παραθέτω μιλάμε, ενώ ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεκάδες εκατομμύρια πρόσφυγες χτυπούν την πόρτα, εκατοντάδες εκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες. Είναι παραπληροφόρηση να λέτε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει υπερασπίζονται τις παράνομες πράξεις των μεταναστών. Είναι παραπληροφόρηση να λέτε ότι η Ευρώπη θέλει να μειώσει τη σημασία τη γλώσσα και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι παραπληροφόρηση το γεγονός ότι οι προτάσεις του Σόρος ε, πάντα ε, στο ίδιο επίπεδο με τις ευρωπαϊκές προτάσεις θέλουν ε, να κρίνονται οι μετανάστες με διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τους Ούγγρους. Αυτά τα πράγματα, σας τα λέω, δεν τα ρωτώ, είναι ερωτήσεις τις οποίες θέτω ε, στην ε, Επιτροπή του Ελσίνκη και στον κύριο Πόλιακ ε, για την ελευθερία των μέσων. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε μία αντιπληροφόρηση που ενημερώνει σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάροκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι καλεσμένη, ακούσαμε με προσοχή τις ομιλίες σας, αλλά ήταν ε, όλες πολύ μονόπλευρες. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ε, εργάζομαι σε μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται και με τη μετανάστευση και έχω πολύ διαφορετική εντύπωση για την κατάσταση που επικρατεί από εσά. Έχουμε πολλά θέματα, εθνική διαβούλευση, διαφάνεια για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπου ε, έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Για, γιατί να μην ρωτάμε τον κόσμο ποια είναι η γνώμη του και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το κάνουμε αυτό και στην Ευρώπη, να ρωτάμε τη γνώμη του λαού. Εγώ, ως ανθρωπολόγος, πιστεύω ότι αυτά που κάνουν οι εμπειρογνώμονες και οι πολιτικοί θύνοντες, ε, έρχονται σε αντίθεση με τη λαϊκή βούληση του κόσμου που μένει στα χωριά, στις πόλεις. Οπότε η διαβούλευση με το λαό, με τη μορφή ενός ψηφίσματος, δεν νομίζω ότι είναι άσκοπη. Επίσης, ε, είπατε ότι μη κυβερνητικέ οργανώσει εξυπηρετούν το λαό. Γιατί λοιπόν να μην γνωρίζει ο λαό από πού χρηματοδοτούνται αυτέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. ούτως ή άλλως για ένα ευρώ από εθνική χρηματοδότηση έχουμε 17 ευρώ από ε, ευρωπαϊκή. Γιατί να μην γνωρίζουμε πώς χρηματοδοτείται κάθε μη κυβερνητική οργάνωση. Και εμείς είχαμε πρόβλημα με τα λογιστικά μας παρόλο που δεν είχαμε ξένη χρηματοδότηση. Το δανεικό και σουηδικό παράδειγμα δείχνουν ότι θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πιο επιστημονικά κριτήρια, πιο ακαδημαϊκά, για να μην έχετε τόσο ε, μεροληπτική άποψη για την Ουγγαρία. Όλες οι διαδικασίες επί που ξεκίνησαν εις βάρος της Ουγγαρίας κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία. Κρίθηκαν ανυπόστατες και αναδαφικές. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι επιδόσεις της Ουγγρικής κυβέρνησης από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Κυρία Παγασάρτον εγώ σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι ξέρω από τον αθνολαϊκισμό, γιατί το βίωσα και στο πετσί μου. Και ένιωσα κι εγώ αυτή την κατηγορία και το στίγμα το αντιφρονούντος. Γιατί το να δέχεται κανείς ε, μία ενιαία ρητορική για το τι εστί εθνική ταυτότητα, αυτό είναι προπαγάνδα. Το να τα την πολιτική, το πολιτικό διάλογο σε, σε συναισθηματικό, αυτό είναι προπαγάνδα, πολύ σοβαρό και μάλιστα δύσκολο καταμετρήσιμο. Γι' αυτό έχουμε και το τέτοιο πρόβλημα. Και καταπατώνται οι αρχές και οι αξίες της πολυφωνίας και του πλουραλισμού. Και μάλιστα οι γονείς του Ιησού της, της, ε, της, του Ναζωρέου ήταν μετανάστες. Ε, και όμως ε, γεννήθηκε από δύο μετανάστες ο Ιησούς Χριστός. Ο κύριος Όλτρα. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα ξεκινήσω με Χριστούς και Χριστούγεννα. Είναι κάπως παράδοξο που είχαμε πάνω από τέσσερις συζητήσεις ε, για την Ουγγαρία και ξεχάσατε ότι δύο φορές συζητήσαμε για τη Ρουμανία. Και από τον Ιούνιο, Ιούλιο και το Σεπτέμβριο μετά εξαφανίστηκε ως διαμαγείας η Ρουμανία. Ενώ η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να εξαφανίζεται από το κατάλογο των συζητήσεων ή τα αντικείμενα της έρευνας. Για να μην αναφέρω τη Μάλτα, την Ισπανία, που δεν παρενοχλούν την κοινωνία υποτίθεται, αλλά απλώς τη πυροβολούν εις βάρος της ή τη φυλακίζουν. ο κύριος Τίμερμας, ο πρώτος αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται να έχασε τον ενθουσιασμό του απέναντι στην έκθεση Ιντβελτ για το μηχανισμό του κράτους δικαίου. Γιατί να μην παρακολουθούμε όλα τα κράτη-μέλη στη συζήτηση και να επικεντρωνόμαστε μόνο σε δύο χώρες, την Πολωνία και τη Ρουγγαρία. Εγώ θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη την έκθεση πρωτοβουλίας και να καταλήξει κάπου. Είδαμε ε, ότι συζητούμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και ξεχνάμε τις υπόλοιπες 25-26 χώρες μέλη. Θα δώσω τώρα με βάση το άρθρο 205 και σε δύο ευρωβουλευτές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Λύπε. Πρώτα στον κύριο Σάνι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Ε, προς τον Υπουργό Εξωτερικών καταρχήν. Η πρώτη ερώτηση είναι γενική πολιτικού χαρακτήρα. Θεωρείτε ότι είναι σωστή η σκέψη της Ουγγρικής κυβέρνησης να επιβάλλει ε, έρευνες σε τέτοιες δραστηριότητες ε, ε, λέγοντας ότι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι εις βάρος ε, της Ουγγαρίας και γίνονται τέτοιοι έλεγχοι στον Ουγγρικό λαό. Επίσης, θεωρώ ότι η αλληλεγγύη έχει πολλές μορφές. Δεν μπορούμε να Ε, ισχυριζόμαστε ότι εφαρμόζουμε αλληλεγγύη παραπλανώντας τον κόσμο. Και αν δείτε τι έγινε με την ε, εκστρατεία για τη διαβούλευση, η βασική ερώτηση ήταν «Θέλετε οι μετανάστες να σκοτώνουν, να βιάζουν τις γυναίκες και τα παιδιά σας» ή να καταπατούν τον πολιτισμό σας. Εάν τεθεί με τέτοιο τρόπο το ερώτημα, φυσικά θα απαντήσουν αρνητικά οι πολίτες. Αλλά δεν είναι αυτό αλληλεγγύη. Ο τρόπος που διατυπώνεται το ερώτημα της λαϊκής διαβούλευσης δεν συνιστά αλληλεγγύη. Επίσης. Κύριε Υπουργέ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε τα τελευταία χρόνια μερικά πολύ αρνητικά σενάρια για τους μετανάστες και έχουμε δεκάδες χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που περιπλανώνται έρημα στην Ευρώπη. 130.000 παιδιά ασυνόδευτοι ανήλικοι θα ήταν δεκτοί ως μετανάστες στην Ουγγαρία. Thank Κύριο Κόμπερν, τελευταίο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ακούω πολλά για τι ευρωπαϊκέ αξίε εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο μέσο του 20ου αιώνα ευρωπαϊκές αξίες ήταν δεξιές, απολυταρχικές, κομμουνιστικές. Γιατί ευρωπαϊκές αξίες μιλάμε. Ουσιαστικά θέλουμε να τονίσουμε τη γραφειοκρατία από ένα μη εκλεγμένο κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως η μόνη δημοκρατική χώρα φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν της αρέσουν ε, οι ευρωπαϊκές αξίες ε, που τις έχουν καθορίσει οι μη εκλεγμένοι γραφειοκρατές. Μήπως θα έπρεπε και η Ουγγαρία να ακολουθήσει το παράδειγμα του Brexit και της Βρετανίας περιμένοντας βέβαια και την αντίστοιχη τιμωρία που μας επιβάλλουν αντιδημοκρατικά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι επειδή τολμάμε να θέλουμε να δικήσουμε τη χώρα μας. Πώς μπορεί, πώς μπορεί λέω, αυτό να είναι ένας ε, δημοκρατικός ε, οργανισμός όταν ε, τιμωρεί τις χώρες που θέλουν να φύγουν και προσπαθεί να κρατήσει τις χώρες δια της βίας. Σύμφωνο Βαρσοβίας μου θυμίζει αυτό, δεν είναι καλή ιδέα. Ελάτε κι εσείς λοιπόν, κάντε τον δικό σας Brexit. It's nice πολύ ωραία κλείσατε την ακρόαση. Ναι, έλεγε και κάτι κάτι ο κύριος διακόπτεται. Διακόπτεται ο κ. Σκόμπερν. Um, uh, Θα ακούσουμε τώρα τη δευτερολογία των ε, προσκεκλημένων μας. Ε, τους ευχαριστώ και τους ζητώ ε, να είναι πειθαρχημένοι. Δύο λεπτά, σίγουρα είναι πολύ λίγος χρόνος και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για ένα τόσο λεπτό θέμα. Απλά είναι λίγο δύσκολο ε, να καλύψουμε το, το χρόνο. Σας ευχαριστώ και εκ των προτέρων για την πειθαρχία. Με τη σειρά που μίλησαν ε, στην πρώτη τους παρέμβαση ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Θα σας δώσω πέντε λεπτά, το πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ουγγαρία θέλει να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε μέλος μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή αν διεξάγει έναν ορθολογικό διάλογο για το μέλλον. Και δεν αφήνει να την κατακλείζει το συνέστημα. Εγώ είμαι 16 χρόνια βουλευτής και το να ακούω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν ε, την ερώτηση αν η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα του μου φαίνεται λίγο περίεργο ερώτημα. Τι ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών σας εξέλεξαν εσάς ε, θα ήταν μια ερώτηση που θα ήθελα να θέσω στην κυρία που με έκανε τώρα ότι τέλος πάντων δεν θα ε, παίξω το ίδιο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε τους Ούγκρους πολίτες και η άποψη αυτή μας καθοδηγεί, ε, είναι ο γνώμονας που διέπει τις δικές μας ενέργειες. Τώρα, η συζήτηση παραλαμβάνω έχει νόημα αν μιλάμε με πραγματικά περιστατικά και γεγονότα και όχι συναισθηματικά φορτισμένα. Όλοι ε, νομίζω με άκουσαν. Δεν νομίζω να είπα ότι όλοι οι μετανάστες είναι τρομοκράτες. Αλλά είπα ότι όταν έχουμε ε, αυτή την ε, άναρχη και παρά τη μετανάστευση με το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων να περνάνε έτσι, ε, μέσα εκεί μπορεί να κρυφτούν πάρα πολύ εύκολα και κάποιοι τρομοκράτες που θα τους στείλουν αυτοί που θέλουν να τους στείλουν σε κάποια μέρη που θα δυσκολεύονται να, να τους στείλουν νωρίτερα. Γι' αυτό και τα δύο τελευταία χρόνια αυξήθηκε η τρομοκρατική απειλή τόσο πολύ σε όλη την Ευρώπη. Και θα αυξηθούν οι μεταναστευτικέ πιέσεις. Συμφωνεί και το ΝΑΤΟ με αυτή τη διαπίστωση. Στη διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Αφρική έδειξε ότι έχουμε Αφρικα, από την Αφρική μεταναστευτική πίεση, η οποία μπορεί να είναι ανεφόρο, ανεφορίων. 60.000 ΜΚΟ, ή τέλο πάντων οργανώσει των πολιτών, υπάρχουν στην Ουγγαρία και ήρθε εδώ και μας μίλησε μόνο. Οι Ουγγροί πολίτες μπορούν να δώσουν το 1% ε, του εισόδηματος στη ΜΚΟ. η ΜΚΟ έχει πάρει δωρές από 282 πολίτες, η οργάνωση που είναι εδώ σήμερα. 700 εκατομμύρια είναι η δημόσια υποστήριξη που παίρνει συνολικά η ΜΚΟ από τον Ουγγρικό προπολογισμό. Η συμμετοχή των ΜΚΟ στην κυβέρνηση ε, και στο κυβερνητικό έργο είναι καλό λέτε, αλλά δεν είναι καλό να γίνονται εθνικές διαβουλεύσεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς που είμαστε στην κυβέρνηση πρέπει και οφείλουμε να ρωτούμε το λαό μας για το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα στρεφόμεθα στον λαό μας για να ζητούμε την άποψή του. Και σε έναν σύγχρονο κόσμο το να θεσπίζονται κανόνες που λένε ότι μία ΜΚΟ πρέπει να δηλώνει την υποστήριξη που λαμβάνει από το εξωτερικό, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι καταπιέζουμε την κοινωνία των πολιτών. Πραγματικό ποιος το ακούσει θα γελάσει, θα του φανεί ηλίθιο, γελίο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι σέβεται η Ουγγαρία όλες τις διεθνείς νόμιες υποχρεώσεις της. Όπως όμως ε, κάνουμε εμείς αυτό, θέλουμε το ίδιο και όποιος έρχεται στην Ουγγαρία να σέβεται το γκρικό δίκαιο. Χορηγούμε το καθεστώς του πρόσφυγα δυνάμει των διεθνών κανονισμών και συνθήκων. Αν κάποιος πλήρει τα κριτήρια, θα λάβει το καθεστώς. Αν όμως δεν πλήρει τα κριτήρια, το αίτημα παροχής ασύλου θα απορριφθεί. υπόθεση Μπάκα κατά Ουγγαρίας. Να σας πω περί πρόκειται. Αν τόσο πια σας φαίνεται σημαντικό. 14 Σεπτεμβρίου 2016 πληρώσαμε αποζημίωση. Εφαρμόσαμε την απόφαση και ενημερώσαμε όλους τους εμπλεκόμενους. Φυσικά Είμαστε στη διάθεσή σας και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θεωρεί ότι κάτι είναι σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί. Μάρτα Παρντάβη τώρα. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αρκετές ερωτήσεις οι οποίες ε, απευθύνθηκαν σε μένα πιο συγκεκριμένα οι αφορούν ε, την πράξη κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, ε, και την κοινωνία των πολιτών στην Ουγγαρία. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, η διαφάνεια είναι σημαντική. Μπορεί να είναι μία καθόλου δικαιολογούμενη αξία και μπορούμε να ρωτάμε και εύλογα ποιος πληρώνει τι στην Ουγγαρία. Οι ουγγρικές μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να συμμορφούνται ε, με την αρχή της διαφάνειας. Πρέπει να αποκαλύπτουμε όλη μας τη χρηματοδότηση, σε τι δαπανώνεται αυτή η χρηματοδότηση, ε, τι δραστηριότητες είχαμε, τι οικονομικές συνέπειες και για την ε, Ουγγρική Επιτροπή του Ελσίνκη. Αυτό συνήθως είναι ένα αρχείο Excel 60 σελίδων, το οποίο γίνεται με ένα πρότυπο το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ε, δικαστηρίου δεν ε, ε, δίνει η Ουγγρική κυβέρνηση ε, οικονομικές λεπτομέρειες. Ε, υποχρεώνει τις ουγγρικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις να ανακοινώνουν από πού λαμβάνουν χρηματοδότηση, ακόμα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε αρκετά θέματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη, ε, την πολιτική και πώς εφαρμόζεται στα θέματα αυτά και πολλά θέματα στον τομέα του ασύλου και της ποινική δικαιοσύνης. Και οι ενισχύσεις που λαμβάνουμε για τα θέματα αυτά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρείται ύποπτη εξωτερική χρηματοδότηση. Υπάρχουν πάρα πολλές ουγγρικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν έχουν όλες ε, πρόβλημα με αυτή την νομοθεσία. Αυτό ακούγεται πολύ συχνά ως επίκριση. Αλλά δεν ε, είναι όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, για θέματα υπεράσπισης πολύ σημαντικών προβλημάτων που διαπιστώνουν κατά την παροχή υπηρεσιών. Και όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, κυρίως ε, τοπική κρατική χρηματοδότηση σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, πρόβλημα, το οποίο δεν επιτρέπει στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να αναφέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, διότι μια κυβερνητική οργάνωση δεν θα λάβει χρηματοδότηση αν μιλήσει για τα προβλήματα. Η χρηματοδότηση από το κράτος έχει και συνέπειες. Ε, Κάποιε ερωτήσει αφορούσαν το άσυλο. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουγγαρία μόλι είπε ότι οι αρχέ εξετάζουν τι αιτήσει ασύλου βάσει ε, του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του πρόσφυγε. Ε, Φέτος ε, στην Ουγγαρία υπάρχουν περίπου χίλια άτομα τα οποία έλαβαν ε, καθεστώς ε, διεθνούς προστασίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους όμως δεν διαμένουν στην Ουγγαρία. Και γιατί αυτό. Βάσει ουγγρικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, κανονικά η Ουγγαρία θα έπρεπε να βοηθήσει και την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμία συνδρομή όμως πέραν της παραμονής ενός μηνών ε, σε ένα καταβλισμό προσφύγων. Από εκεί και πέρα ε, βρίσκονται αντιμετώπιοι με τη φτώχεια και την εξαθλίαση και την ε, τεράστιο ρατσισμό τον οποίο υποδαβλίζει η κυβέρνηση. Οι προσφύγες λοιπόν υποχρεούνται να μετακινηθούν και να πάνε αλλού και φεύγουν φυσικά. Τον Απρίλιο φέτος Βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου αποφασίστηκε να μην επιστρέφονται οι αιτούντε άσυλο στην Ουγγαρία και έτσι ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία δυνατότητα προστασίας για αυτούς τους πρόσφυγες, όχι γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα, και πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τους κρατήσουν εκτός χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γκάμπορ Πόλεκ για πέντε λεπτά επίσης. Σας ευχαριστώ. Ίσως ναι. σήμερα δημιουργήσετε την εντύπωση ότι η συζήτηση σήμερα δεν αφορά τα μίντια. Ε, εγώ διαφωνώ. Ε, η κατάσταση για τη μετανάστευση ίσως εν μέρη παρουσιάστηκε με τόσο παραπλανητικό τρόπο λόγω της ε, μονομέρειας και των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης γιατί ο πληθυσμός έχει περισσότερο πρόσβαση στα προπαγανδιστικά κυβερνητικά μηνύματα και είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς μια ε, εχθρική εκστρατεία μέσω των κρατικών μέσων. Οποιοςδήποτε όμως ξεκινήσει μια εχθρική εξτρατεία κατά της κυβέρνησης θα στιγματιστεί ως υποχείριο του Σόρος, μισθοφόρος του Σόρος ή κάτι χειρότερο ακόμη. Αυτό συμβαίνει μέσω των ΜΜΕ που τα τελευταία χρόνια έχουν υποταχθεί ή υπαχθεί στον κυβερνητικό έλεγχο. Στην περίπτωση των ΜΜΕ Έχουμε μια πολύ απλή κατάσταση και πολλούς δείκτες. Freedom House, δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Έχουμε εκθέσεις που ε, δημοσιεύονται ετησίως, είναι προσιτές σε όλους και καταμετρούν αυτή την κατάσταση στα ΜΜΕ. Όλες λοιπόν οι οργανώσεις με τον ΑΒ τρόπο χαρακτηρίζονται από το ΦΙΔΕΣ ως ε, ε, πιόνια μιας συνωμοσίας μιας πλεκτάνης που έχει ξεκινήσει ο όρος. Αυτή είναι η, απλο, η απλουστευμένη εντύπωση που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση. Επίσης, αν αφισβητείτε την ελευθεροτυπία, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν απολυθεί από τοπικές εφημερίδες, από τοπικούς ή κρατικούς ραδιοτηλεπτικούς σταθμούς. Χρειάστηκε να αλλάξουν επάγγελμα και μια πολύτιμη κρίσιμη μάζα δημοσιογραφική χάθηκε ε, στα ΜΜΕ λόγω της πολιτικής επέμβασης που έχει πλήξει όλα τα επίπεδα των μίντια. Επαναλαμβάνω, πολλοί δημοσιογράφοι άλλαξαν επάγγελμα και όσοι έμειναν είναι υποχρεωμένοι να παίξουν το παιχνίδι της κυβέρνησης και να εξυπηρετούν τις επικοινωνιακές ε, ανάγκες της κυβέρνησης. Κάποιο είπε ότι η εκστρατεία εθνική διαβούλευση είναι καλό μέσο ε, διαβούλευση με του πολίτε. Εγώ δεν έχω διαβάσει τέτοιο ερωτηματολόγιο και άσχετα από την παράταξη την ε, πολιτική του καθενό. βλέπει τι παγίδα είναι αυτή η εθνική διαβούλευση. Τα ερωτήματα δεν είναι πραγματικά ουσιαστικά ερωτήματα και άμα δεν έχουμε ουσιαστικά ερωτήματα πώ περιμένετε πραγματικές ε, ουσιαστικές απαντήσεις. Η μόνη ουσιαστική απάντηση είναι ότι Ό,τι και να απαντήσετε θα ενισχυθεί θέση του Φίδες. Το Φίδες θα χειραγωγήσει απαντήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ευλογήσει τα γένια του. Ούτως ή άλλως τα ερωτηματολόγια δεν καταχωρούνται καν, οι απαντήσεις δεν καταχωρούνται καν, δεν, δεν πρόκειται για ουσιαστική συζήτηση, δεν πρόκειται για διάλογο εθνικό. Επίσης κάποιος ρώτησε τι συνέβαινε πριν το 2010. Σας ε, λέω ειλικρινά ότι α, δεν ε, θα διαβάσετε κανένα δικό μου άρθρο τότε που ε, επενούσε το, τα μίντια πριν την κυβέρνηση Φίντες. Υπήρχαν ομάδες λόμπι, υπήρχε κυβερνητική επιρροή αλλά αυτή η κατανομή των κρατικών ενισχύσεων ε, ήταν πολύ πιο δίκαιη πριν το 2010, παρά τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα. Είχαμε κρατική παρουσία στις ε, διαφημιστικές εκστρατείες, αλλά όχι τόσο μαζική όσο σήμερα. Σε μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 100% των εσόδων προέρχονται από το κράτος. Και εγώ θέλω να ζω σε μια χώρα που είναι ελεύθερη, όχι μόνο λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ζω σε μια χώρα που θα υπάρχει ελευθεροτυπία, που δεν θα νιώθω στο στόχαστρο των επιθέσεων. Και αυτό δεν το λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέω για την Ουγγαρία, για τα παιδιά μου, για του φοιτητέ μου, για του συμπολίτε μου. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη και μακάρι να το κάνει, αλλά όλα αυτά που κάνω δεν τα κάνω για την Ευρώπη, αλλά για την πατρίδα μου την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Σάντο για πέντε λεπτά επίσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στην Ουγγαρία που θα πίστευε πραγματικά ότι είναι σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. ή ότι χρειάζεται ε, αποκατάσταση του κράτους δικαίου. δεν βλέπω κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες. Ε, προς απάντηση στην κυρία Αργεντινή, κοίταξε κοίταξα το άρθρο 2, που οι ορισμοί είναι σαφείς. Μιλάμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ε, ισότητα, κράτος δικαίου, πλουραλισμός, δικαιώματα καταπολέμηση διακρίσεων, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα είναι ξεκάθαρη σε αυτές οι έννοιες. Ο καθένας μπορεί να τις ε, εννοήσει όπως ε, νομίζει. Είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι οικουμενικές αξίες. Ποιο είναι το βασικό δικαίωμα για έναν ε, ε, μετανάστη να πάρει ε, άσυλο ε, στην πρώτη ασφαλή χώρα ή οπουδήποτε θέλει. Τι θα γίνει, παραδείγματος με τους γάμους ομοφιλοφίλων. Σε πολλές χώρες της Ένωσης δεν είναι νόμιμη αυτή η γάμη. Άλλα συνταγματικά δικαστήρια λένε όμως ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα και ανθρώπινο δικαίωμα γάμος μεταξύ ομοφιλοφίλων. Και το κράτος επίσης πρέπει να αναγνωρίσει άλλα φύλλα ε, πέραν των δύο που έπλασε ο Θεός. Άλλοι, ε, άλλα κράτη δεν το δέχονται αυτό. Υπάρχει δυνατότητα προστασίας και πρόσπισης της ε, Ιουδοχριστιανικής παράδοσης που είναι η πλειοψηφία στη Γαλλία. Μήπως κατεβαίνουν οι σταυροί γιατί δε, σε κάποιους δεν αρέσει αυτό το σύμβολο. Η προστασία της ζωής του εμβρίου. Σε κάποιες χώρες υπάρχει επιλογή ε, άμβλωσης, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει. Ωραία λοιπόν να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και να λέμε όλες αυτές τις λέξεις, αλλά είναι ασαφείς οι ορισμοί, είναι αφηρημένες οι έννοιες. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο ο καθένας να γεμίσει, αν θέλετε, ε, τις ε, ε, λέξεις με το νόημα που επιθυμεί, τροπή Βενετίας, αρχαία τα κτλ. Τι γίνεται λοιπόν με το κράτος δικαίου τι γίνεται όταν σε ένα κράτος έχουμε εντοπίσει πρόβλημα, κράτος δικαίου. Λέτε περικοπή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία, η κεντρική Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, έχει πολύ τραυματικό παρελθόν. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πιάσαμε αν θέλετε το Μουτζούρι εμείς. Το ίδιο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθαν οι Ρώσοι. Μετά τις αλλαγές, μετά το 1989 και πριν το 2004, απελευθερώσαμε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, της αγορές μας, με τα ακολούθηση προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίξαμε τις αγορές μας όπως και την αγορά εργασίας βλέπετε ότι υπάρχει κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και επίσης συνεισφέραμε και στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας. Μην αρχίσετε να μου λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά οι Βρυξέλλες μας ε, κάνουν ε, ελεημοσύνη και μας τα προσφέρουν όλα. Κάναμε πάρα πολλά για να είμαστε επιλέξιμοι για αυτή την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. και τις προϋποθέσεις και τους όρους που επιβάλλουν ε, από την Ένωση για να μας δίνουν αυτή τη του τους στηρούμε. Πρόεδρος. Από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι έρχονται για την ψηφοφορία, θα ολοκληρώσουμε τόσο λίγο. Οι σκιώδει συγητέ θα συζητήσουν, θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτή τη ακρόαση. Να ευχαριστήσω του σκιώδει συγητέ και την εισηγήτρια για το δουλειά του σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Σα παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγο ησυχία μέχρι να ολοκληρώσουμε. Ε, το σχέδιο έκθεσης θα παρουσιαστεί το Μάρτιο, θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό και ε, θα δώσω στην εισηγήτρια ε, το λόγο για δύο λεπτά για να κάνει τις τελικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι στιγμή για συμπεράσματα ακόμα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο και αργότερα στο Σεπτέμβριο. Επομένως είναι πάρα πολύ πρόημο να καταλήξω σε συμπεράσματα. Θα ήθελα απλώς ε, να κάνω δύο παρατηρήσεις ολοκληρώνοντας. Όπως είπα προηγουμένως, ε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 που εξηγεί ότι η διαδικασία για το άρθρο 7 είναι κάτι παραπάνω από κάποιες ε, διαδικασίες επί παραβάση. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Μπορεί οι διαδικασίες επί παραβάση είναι ε, σημαντικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Τα θέματα είναι επιτάπητος και πρέπει να ε, καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας πάρα πολύ προσεκτικά. Το άλλο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω και στο οποίο νομίζω αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική να μην ε, ε, ε, αναμειγνύουμε κράτος, κυβέρνηση, κόμμα και λαό. Ένα κόμμα δεν είναι κυβέρνηση, ένα κράτος δεν είναι κυβέρνηση ή κόμμα και οι άνθρωποι είναι μεμονωμένα άτομα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να συμφωνήσω με κάποιον που είπε ότι εμείς δεν κοιτάμε και δεν κρίνουμε την Ουγγαρία. Εμείς είμαστε με τη χώρα, με την Ουγγαρία και εξετάζουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και την κατάσταση στην Ουγγαρία προς όφελος ε, των Ευρωπαίων και Ούγγρων. Ε, ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνέχεια της ε, συνεργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητέ και τα μέλη. Ήταν πολύ ευαίσθητα τα πολιτικά θέματα αυτά σε μια πάρα πολύ ε, περιορισμένη κατάσταση. Ευχαριστώ όλους για την πειθαρχία τους και να ευχαριστήσω και τους παρισταμένους για την ακρόαση. Η ακρόαση ολοκληρώνεται. Η έκθεση θα εκπονηθεί το Μάρτιο. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα διακόψω για 30 δευτερόλεπτα ε, για να βιάσει το Προεδρείο. As a colleague, just prepare for the vote. I know we have to go quickly because people will have to leave. I realise this. Stay where you are if you're voting. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Σας παρακαλώ ε, να είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Thank you. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Καθίστε, παρακαλώ. Αν δεν σκοπεύετε να συμμετέχετε στην ε, ε, ψηφοφορία, Ψηφίζουμε λοιπόν ε, ε, το, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την επιχειρησιακή διαχείριση μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης. Ε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μακοβέη. Κυρία Μακοβέη, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία. Την κυρία Κινίτσι το ΕΠΠ, e το ΕΛΚ και τους υπολείπους και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά σύντομα και ακούσαμε και τις τεχνικές εξηγήσεις των εμπειρογνωμόνων. Επομένως, ε, θεωρώ ότι όλα πήγαν πολύ καλά ε, και πήγει το ζήτημα, διότι ασχολούμαστε με το EU LISA, την διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, τη συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει υποχρέωση γι' αυτό και το επισημαίνουμε και την καταπολέμηση ε, ε του τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της προκλήσης της μετανάστευσης, τις οποίες θα μπορούσαμε να επιλύσουμε εν μέρη, εάν έχουμε ένα σύστημα υγιουλίσσα που να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κύριε Μακοβέη. Κύριε Βίξτρομ, έχετε κάτι διαδικαστικό. Ναι κύριε Πρόεδρε, έχω κάτι διαδικαστικό. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα να ζητήσω επικαιροποίηση της ε, ε, του καταλόγου ε, ψηφοφορίας βάσει του άρθρου 195 του κανονισμού και να σας εξηγήσω γιατί. Προτείναμε να υπάρχει επικαιροποίηση μέχρι τουλάχιστον τις 15 Ιανουαρίου και ε, ο λόγος είναι ο εξής. Εδώ πρόκειται για νομοθεσία που είναι πάρα πολύ σημαντική διότι ε, η Ιουλίσα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για την ε, παροχή μακροπρόθεσμων λύσεων για την επιχειρησιακή διαχείριση ε, πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Αυτό σίγουρα θα έχει τεράστιες συνέπειες για την αρχιτεκτονική δομή των θυσιμάτων, την ασφάλεια και τη δημοκρατική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη ε, ως διαπραγματευτική, διότι η διαπραγματευτική διαδικασία εδώ στο Κοινοβούλιο ήταν ε, ε, βεβαιασμένη και δεν ήταν και κατάλληλα δομημένη. Η πρόταση ε, κατατέθηκε τον Ιούνιο. Η διαπραγμάτευση της έκθεσης έγινε για δύο εβδομάδες μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο. Δύο μόνο εβδομάδες, δύο πολύ σύντομες συναντήσεις σκιωδών εισηγητών και αυτό πρέπει να το δείτε σε αντιπαράθεση με άλλα νομοθετικά θέματα. 22 συναντήσεις των σκιωδών μέχρι να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο, η, η, συγγήτρια δεν ε, ε, δέχτηκε να ε, καλωσορίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΛΚ ε, και ε, άλλου στην ε, ε, συνεδριάση των εισηγητών, παρά το γεγονό ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, θα μπορούσαμε να είχαμε εξηγήσει μεταξύ των διαφόρων φορείων. Συνολικά ήταν μια βεβαιασμένη διαδικασία, την οποία πιέσαμε πάρα πολύ πρόημα, πιστεύω. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει μια πολύ ισχυρή εντολή για το Ιγιουλίσα. Διότι ανοίγουν οι θύρε για την διαλειτουργικότητα με αυτόν τον τρόπο και γνωρίζουμε όλοι ότι η πρόταση αυτή προέρχεται θα, μάλλον θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρακολύσω τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει η διαδικασία να γίνει με σωστό τρόπο, με τη σωστή νομική βάση και δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εάν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία σήμερα, σίγουρα θα καταψηφίσουμε είναι διαδικαστικό βάσει του άρθρου 190 παράγραφος 4, το αναφέρατε. Αυτό το άρθρο προβλέπει η πλειοψηφία των παρισταμένων να πούν αμέσως πριν από την ψηφοφορία κατά πόσον θα πρέπει να διακοπεί η ψηφοφορία. Ε, κυρία Μακοβέη, θέλετε το λόγο? Και να τονίσω το εξής πριν λάβετε το λόγο. Συνάδελφοι σας, παρακαλώ λίγο ησυχία. Δεν θέλουμε να ξεκινήσει εδώ συζήτηση, διότι ε, στο διαδικαστικό θέμα ε, μπορεί να μακρηγόρησε λίγο η ομιλήτρια μεν, αλλά ζητά διακοπή της ψηφοφορίας. Ε, και ξέρω ότι οι συνάδελφοι θα θέλουν να ψηφίσουμε ε, γρήγορα. Η κυρία Γουίξτρομ εξήγησε πάρα πολύ καλά τι θέλει. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να διακοπεί ψηφοφορία βάσει του άρθρου 190 παράγραφος 4, το οποίο προϋποθέτει άμεση ψηφοφορία και απαιτεί πλειοψηφία των παρισταμένων. Θα ήθελα λοιπόν να ψηφίσουμε απευθείας για να δούμε αν θα γίνει ψηφοφορία ή όχι. Θέλετε να ξεκινήσετε συζήτηση, κυρία Μακοβέ, γιατί φαντάζομαι ότι θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά, το αντιλαμβάνομαι. Θέλετε να απαντήσετε πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Παρά το διαδικαστικό, το οποίο δεν είναι διαδικαστικό, θα είμαι πολύ σύντομα. Έγινε μια τεχνική συνεδρίαση με το EDPS και το EULISA κατόπιν αιτήματος των φιλελευθέρων. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε συνεδρίαση Όλοι οι υπόλοιποι σκιώδει ηγητέ ε, αρνήθηκαν να συμμετέχουν διότι είπαν είμαστε πεπισμένοι, δεν το χρειαζόμουν και οργανώσαμε τη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο κατόπιν αιτήματο τη κυρία Βίξτρομ. Και εκπλήσωμε που οι δύο, σκιώδεις, ε, ε, οι δύο συναντήσεις με τους σκιώδεις συζητητές ήταν πάρα πολύ καλές. Βρήκαμε συμβαστικές λύσεις σε όλα, εκτός από ένα σημείο. Και είμαι εντελώς αντίθετη σε αυτό. Ευχαριστώ. Εκτιμώ μας το επισημάνατε και μιλήσατε και τις ε, συνεδριές των σχεδιών. σχεδίων. Ήταν όμως γνήσιο διαδικαστικό της κυρίας ε, Wickstrom γιατί επικαλέστηκε συγκεκριμένο άρθρο και υπέβαλε το διαδικαστικό με βάση αυτό το άρθρο. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Μπορούμε να ψηφίσουμε διανατάσσεως της χειρός ή θέλετε μήπως ηλεκτρονικά. Όχι, όλα ηλεκτρονικά τα κάνουμε στην Επιτροπή μας, οπότε ψηφίζουμε, παρακαλώ. και λίγη ησυχία παρακαλώ. Αν ψηφίσετε πράσινο, υπέρ δηλαδή, σημαίνει ότι θέλετε να γίνει ψηφοφορία. Αν ψηφίσετε κόκκινο, κατά, σημαίνει ότι δεν θέλετε να γίνει ψηφοφορία του θέματος της έκθεσης αυτής. My uh, συγγνώμη, δίκιο έχει η κυρία Χολμάιερ. Σας μπέρδεψα χειρότερα, σας απογοήτευσα και ζητώ συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να επανορθώσω. Λοιπόν, θα ψηφίσετε ναι, πράσινο, αν θέλετε αναβολή της ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Όποιος θέλει να αναβάλουμε την ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσει ναι και όχι αν είναι κατά της αναβολής. Ψηφίσετε ναι αν είστε υπέρ της αναβολής και όχι αν είστε κατά της αναβολής. Και ρίξτε και μια ματιά στους συντονιστές σας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο έξυπνο συγκεκριμένη περίπτωση. Κυρία Χολμάγερ, δεν έβαλα ακόμα την κάρτα. Εγώ να, δείτε πώς έχω απογοητευτεί, κυρία Χολμάγερ, από εσάς. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας, οπότε το αίτημα της αναβολής απορρίπτεται και άρα θα ψηφίσουμε. Δεν έχουμε πια ουγγρική διερμηνία γιατί η ουγγρική καμπίνα πήγε στη συνέντευξη τύπου. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 7. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 83 με 85 μαζί. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 86, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 88, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Άρχεται η ψηφοφορία. 92. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της Επιτροπής Προπολογισμών. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 102 με 104 μαζί. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Συμβαστική 4. η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 με, μέχρι 111 μαζί, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνονται. 113, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 114, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέσσερα της Επιτροπής Προπολογισμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Εγκρίνεται. Συμβαστική, πε... Ε, μάλλον τροπολογία 5 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6, άρχεται η ψηφοφορία. Α, πρέπει να πω με ονομαστική κλίση. Πρέπει να ακουστεί αυτό πρώτα. Οπότε για τη συμβαστική έξι ονομαστική ψηφοφορία. Αν δεν το πω φωναχτά, δεν θα καταγράφει έτσι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε 117 με 119 μαζί, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. 63 μέχρι 65 άρχεται ψηφοφορία. 63, 64, 65. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Προϋπολογισμών, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 126, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 20 Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 131. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 132 και 133 μαζί. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. 134. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 135. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 136 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 26 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 8 της Επιτροπής Προϋπολογισμών άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 29. Άκτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άκτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 31. Άκτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 32. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 33 και 144 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται. 147 έχετε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 148 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 150 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 151 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 152 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 153 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 155. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 156. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 157 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 158 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 159 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 37-160 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 161 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 38 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Προϋπολογισμοί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 162 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 163 έχετε ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 164 πρώτο τμήμα η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα 164 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκτό και αυτό. Πάμε στην τροπή 40. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική όχι. Λάθος. 165. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 42 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 12 προϋπολογισμή άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 171 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 44 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προπολογία 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 15. Άρχισε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 16 προπολογισμοί. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται 17 προπολογισμένα έρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 15 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 50 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 51 υπέρ. Μάλλον άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Κλωτσάει κανεί το έδρανό του. Κάπως με αποσυντονίζει. Ε, με, είναι εντάξει, αγχωτικό. Μου έρχεται και εγώ να αρχίσω να κλωτσάω, δεν πάντων. 176 άρχεται η ψηφοφορία. Και πολλά μπορώ να αρχίσω κοπανάω, αλλά τέλο πάντων. Άρχεται η ψηφοφορία το 176. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε σε λογικές αναφορές. 54. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 72 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 73 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 74 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 75 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 προπολογισμοί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 4 αποχές. Και τώρα θα ψηφίσουμε την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 40 υπέρ, 11 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εδώ ολοκληρώθηκε η ώρα ψηφοφορία αγαπητοί συνάδελφοι. Συνάδελφοι, όσοι από εσά θα παραμείνετε, πάμε απευθεία στο σημείο 8. Αν σκοπεύετε λοιπόν να παραμείνετε, σας παρακαλώ ε, ήσυχα και όσοι φεύγετε αποχωρείτε ήσύχο παρακαλώ. Και πάμε απευθεία στο σημείο 8. Είναι θέμα της κυρίας Έρνστ. Ε, Η Κορνίλια Έρνστ είναι εδώ. Ah. Sorry, Uh, Mrs. I didn't see you. Uh, Συγγνώμη, κυρία Έρνστ, δεν σα είδα. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ ε, λίγο ησυχία, διότι έχουμε δύο ακόμα θέματα στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα ε, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Παρουσίαση λοιπόν της κατάστασης ε, για τις διαπραγματεύσεις και τον τριμερή διάλογο για την προστασία ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα θεσμικά όργανα, φορείς, γραφεία και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Η εισηγήτρια είναι η Κορνίλια Ένστ και πάλι όπως και με πολλούς άλλους τριμερείς διαλόγους υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ όλους εκείνους που εργάζονται πολύ σκληρά για διάφορους τριμερείς διαλόγους. Ένας εξ αυτών είναι ο συγκεκριμένο και μετά την έγκριση της ε, ε, έκθεσης Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στις 9 Οκτωβρίου, η κυρία Ένστ ξεκίνησε το διάλογο και θα της δώσω το λόγο για να μας κάνει μια ενημέρωση. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. <laughs> Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich möchte... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για το έχει κατάσταση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο στόχος ε, του κανονισμού ήταν και είναι ε, η εφαρμογή ε, του νέου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένους τομείς. Θα πρέπει ακριβώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εφαρμόσουμε αυτό το καθεστώς. Αυτό σημαίνει και για τους οργανισμούς και διάφορους φορείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, υπάρχει πολυσχηδής κατάσταση και γι' αυτό ε, υπάρχει αυτή η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς έχουν όμως τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, ε, ζητήματα μάλλον, των οποίων καταφέραμε να βρούμε πολύ γρήγορα ε, συμβιβαστικές προτάσεις ε, και να καταλήξουμε σε συμφωνία χθες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδαμε τα ανοιχτά σημαντικά ζητήματα και μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις. Αλλά δεν έχουμε κλείσει με όλα τα θέματα. Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση, δεν είναι διατεθειμένο να συζητήσει σοβαρά τα ζητήματα αυτά. Ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι τα βασικά ζητήματα, τα ανοιχτά ζητήματα, το scope πρώτα απ' όλα, το δεν εφαρμογή. Δεν μπορούμε από αυτό το scope ε, ξαφνικά οργανισμούς, άλλους φορείς ε, να σου βγάλουμε και να πούμε ότι για αυτούς δεν ισχύουν αλλά ε, γενικά τα άλλα πρέπει να ισχύουν. Όχι, για τη Europol, τη Eurojust και το γραφείο του ε, εισαγγελέα θεωρούμε ότι στο σκοπ πρέπει να συμπεριληφθούν και σε ό,τι αφορά την αρμόνιση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όχι να εξαιρεθούν. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για κάτι τέτοιο. Ως κοινοβούλιο κάναμε τις προτάσεις μας γιατί θέλουμε το συμβιβασμό προτείναμε για τη Europol παραδείγματο χάρη να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και ενδεχομένω ε, τα προβλήματα που μπορεί τώρα, εμεί να μην τα βλέπουμε, αλλά τέλο πάντων, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, ε, να υπάρχει η δυνατότητα μετά από αυτή τη μεταβατική περίοδο να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση. Αυτή είναι η πρώτη πράξη που μπορεί κανείς να διατυπώσει. Για το Συμβούλιο λέει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αρμόνιση των ε, δικαιωμάτων των ε, προσωπικών μάλλον δεδομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την ε, Eurojust, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και στο πλαίσιο αυτού κανονισμού. Από ό,τι φαίνεται, Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ε, να βάλουμε κάποια πράγματα τα οποία μετά θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Δεν ε, υπάρχει κάποια αιτιολόγηση ούτε εδώ. Ούτε εδώ το Συμβούλιο ήθελε να μας πει συγκεκριμένα όπως για την Europol, έτσι και για την Eurojust, να μας πει γιατί προτείνει αυτά που προτείνει, για τη Eurodac εντάξει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί θα ενταχθεί στο ΛΙΣΑ, στο EU ΛΙΣΑ, το Eurodac. Δεν είχαμε εκεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Για το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, όπως και για τη Europol, έχουμε την ίδια άποψη. Νομίζω ότι μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία, δηλαδή με την θέσπιση μιας μεταβατικής περίοδου, αν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα, αλλά στη ζωή μας πρέπει να αναζητούμε συμβιβασμούς και εμείς είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, συζητήσουμε τις ε, αποστολές του δεύτερου πυλώνα ιδίω ε, που δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, όπως πάντοτε είμαστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για το κεφάλαιο 8α δεν είμαστε ευέλικτοι. Δεν θέλουμε να το θάψουμε, διότι θεωρούμε ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε επίσης ότι είναι παράλογο να πούμε ότι για άλλες νέες ε, ε, agencies και τα λοιπά, ναι. ναι. να ισχύει αυτό, αλλά όχι για την Europol, όχι για την Eurojust και όχι για το γραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ε, δυνατή αιτιολόγηση, ούτε λογική εξήγηση. Αυτά είναι τα ανοιχτά προβλήματα. Και κάτι άλλο. Για του εσωτερικού κανόνε νομίζω ότι εδώ έχουμε δυνατότητα να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Και αν είχαμε ολοκληρώσει τα προηγούμενα θέματα που σα ανέφερα, θα είχαμε τελειώσει και με αυτό, θα είχαμε καταλήξει σε μια καλή λύση και θα μπορούσαμε να τα αποφασίσουμε όλα την επόμενη εβδομάδα. Εγώ πρέπει να πω ολοκληρώνοντα ότι το Συμβούλιο δεν εκπληρώνει το καθήκον του, δεν εργάζεται μαζί μα ε, με ειλικρίνεια και με σοβαρότητα ε, σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των ε, στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα. Είμαι πολύ απογοητευμένη με το Συμβούλιο και πραγματικά είμαι απογοητευμένη. Ε, δεν ξέρω πού μπορούμε να βασιστούμε. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά ζητάμε ε, το Συμβούλιο να ασχοληθεί για αυτά τα τρία οργανισμούς που είπα ε, πολύ σοβαρά μαζί μας και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δεν ήταν διατεθειμένοι για κάτι τέτοιο. Η ευθύνη ανήκει στη πλευρά του Συμβουλίου. Δεν έχει αναλάβει ακόμη τις ευθύνες του Οι προηγούμενε προεδρίες κάναν ό,τι μπορούσαν. Ε, το σέβομαι ε, και θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία και τους σκιώδεις βέβαια πάνω απ' όλα, οι οποίοι ε, μου έδωσαν κουράγιο και με παρότερα να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τη γραμματεία της Λίμπε αλλά ούτε και την Κομισιόν που ευτυχώς ε, δείχνει λογική και μας βοηθάει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ένστ. Προσπάθησα λίγο να παρακολουθήσω το θέμα και νομίζω ότι είναι καλό για τα μέλη να ακούσουν γιατί υπάρχουν προβλήματα και ε, για όσους ε, δεν είναι εδώ να ακούσουν τα καλά σας λόγια. Ε, η αίσθησή μου είναι ότι η Εσθενική Προεδρία πρέπει τώρα να παραδώσει το θέμα στη Βουλγαρική Προεδρία. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε πλέον. Καλό είναι όμως να ξέρουν και τα μέλη της Επιτροπής μας γιατί είναι τόσο απογοητευτική η κατάσταση. Ναι, δεν είπα τίποτα ουσίας, μην ανησυχείτε. Ε, ευχαριστώ και πάλι για την ε, έκθεσή σας. Συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει κάποιος ε, Γιάννη, εσύ παρακολουθείς το θέμα, θέλεις να πεις κάτι, ο κύριος Άλμπρεχτ. Θα ήθελα απλώς ε, να ευχαριστήσω την Κόνη για τη δουλειά της στις διαπραγματεύσεις και να συμφωνήσω με την ανάγκη τα κράτη-μέλη να ε, προχωρήσουν για το αίτημά μας να έχουμε ένα αρμονισμένο πεδίο εφαρμογή για τους βασικούς τομείς. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι θέλουμε να επιτύχουμε διαλειτουργικότητα και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών στο τομέα της επιβολής του νόμου και δεν είναι λογικό να έχουμε κοινά πρότυπα για τις αρχές των κρατών μελών μόνον. Ε, προφανώς ε, θα πρέπει να έχουμε και κοινά πρότυπα και ορισμούς για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα συστήματά τους, ε, ιδάλλως δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι διατάξεις και οι ορισμοί και θα ήταν κρίμα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ, Γιάν. Ε, θέλετε να πείτε και εσείς δύο λόγια. Ευχαριστώ. Πολύ απογοητευτικά όλα αυτά. Ούτε και εγώ καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αποκλείουμε τη Europol και τη Eurojust από το κοινό σύστημα. Δεν το κατάλαβε ότι κάνει ηγήτρια. Οπότε φαντάζεστε γιατί γίνεται αυτός ο αποκλεισμό. Είναι θέμα ασφάλεια μόνο. Και άρα εμπίπτει στην εθνική κυριαρχία με βάση και τις συνθήκες ή υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος που κρύβεται πίσω από αυτόν τον αποκλεισμό. Θα μπορούσατε να πιθανολογήσετε ενδεχομένω. Δεν χρειάζεται τώρα, Κόνη, άμα δεν θες να ξεκινήσουμε συζήτηση. Όντως πάντως ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θέλεις να το σχολιάσεις. Είναι πολύ απλό αν δει κανείς τα κρατάμε τη μέλη, τι γίνεται, αυτά οι κανόνες ισχύουν ουσιαστικά ε, και θα έπρεπε αυτές οι προϋποθέσεις ε, να εφαρμόζονται. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, θα έπρεπε να μπορεί να ισχύει. Για την Ευρωπόλ δεν ξέρω. Ούτε καν για ποιους λόγους. αλλά έχει γίνει και με μεταρρύθμιση του ε, κανονισμού. Εγώ δεν βλέπω καμία λογική εξήγηση. Καλώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κόνη, για την ενημέρωση. Και τι να σου πω, καλή τύχη με την Βουλγαρική Προεδρία. Εμεί θα σα στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Και περνάμε στο σημείο 9 τώρα. Μία σύντομη ενημέρωση για την αποστολή μας στην Βόσιγκτο. Γιατί τους άλλους έχουν εξαφανιστεί οι συνάδελφοι από την αίθουσα. Πρόκειται για την αποστολή, την ad hoc αποστολή που πραγματοποιήσαμε 17 ε, με 21 Ιουλίου τρέχοντος έτους στην Ουάσιγκτον. Σαν πέρασε αιώνα από τότε. Πολύ σημαντική πάντως ε, και αποτελεσματική η αποστολή μας. Να και έχουμε μείνει τρεις και ο Κούκος, βέβαια η κυρία Τσινίτσι είναι παρούσα. Ε, και το προσωπικό υπάλληλοι μας φυσικά είναι εδώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Πάντως ήταν σημαντική η αντιπροσωπεία. Εφτά συνάδελφοι από τη Λίμπε μαζί με την κυρία Τζινίκη. Ευχαριστούμε που αν μη τι άλλο εσείς δίνετε το παρόν κυρία Τσινίκη και επαληθεύετε και αυτά που λέω. Εφτά λοιπόν ήταν οι συνάδελφοι, εφτά μελής αντιπροσωπεία και ο υποφαινόμενος μετέβησαν στη Ουάσιγκτον να κάνω μια σύνοψη των πεπραγμένων. Πάντως ήταν πολύ καλά στοχευμένη και εστιασμένη η αντιπροσωπεία μας σε θέματα ύψης της σημασίας, προστασία των δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητα, η Αμερικανική Ασπίδα της Ιδιωτικότητα, λίγο πριν την κοινή αξιολόγηση, η Γενική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για την κρυπτογράφηση, επιβολή του νόμου, ουδετερότητα του δικτύου, αντι, αντιτρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση, ξένοι μαχητές και ούτω καθεξής πολύ σημαντικό θέμα το πρόγραμμα των ΗΠΑ για την εξαίρεση από τις θεωρίες και την αμοιβαιότητα. Όλα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θα μπορούσα να, να μιλώ πολλή ώρα για όλα αυτά, αλλά μια και δεν υπάρχει ακροατήριο για να έχουμε συζήτηση. Α, ήρθε και η κυρία Μπεσερίλ. Σας ευχαριστώ. Δύο καταπληκτικά εκλεκτότατα μέλη της αντιπροσωπείας ε, παρέμενα στην αίθουσα. Και εσύ βέβαια κόνησε εδώ ακόμη, αλλά δεν ήσουν στην ε, Επιτροπή της Λίμπης στην Βόσικτον. Εν πάση περιπτώσει. Ε, θεωρώ ότι δείξαμε τον καλύτερο μας σε αυτό και πραγματικά πρωτοστατήσαμε στη συζήτηση πολύ σημαντικών θεμάτων και παρόλο που πέσαμε σε μια μεταβατική περίοδο, όχι μόνο πολιτικής μετάβασης, αλλά και μετάβασης διοικητικής, αλλαγή ε, διοικητικού προσωπικού και πολλοί ένιωσαν ότι δεν θα έχει και μεγάλη βαρύτητα η αποστολή, αλλά ακριβώ επειδή επικεντρωθήκαμε σε πολύ σημαντικά θέματα ιδιωτικότητα, ε, εξαίρεση από τι θεωρήσεις και ούτω καθεξής, πολύ σημαντικά θέματα, αντιτρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση, θύματα και ούτω καθεξής. Και ακριβώς λόγω της προσήλωση και της δέσμευση των μελών της Επιτροπής και λόγω της πολύ καλής άρτια διοργάνωση του προγράμματος, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου εκτίμηση. Και πραγματικά για μένα ήταν μεγάλη χαρά αυτή η αυτό το κοινό ταξίδι με τα μέλη των, ε, της αντιπροσωπείας. και σε άλλα ταξίδια πω, και μπορώ να κρίνω ότι το συγκεκριμένο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και πολύ καλή επαφή και επικοινωνία μεταξύ μας. Καταφέραμε και διεκπαιρώσαμε και ερευνητικό έργο σε ό,τι αφορά την Αμερικανική Ασπίδα Ιδιωτικότητα και την ε, επικείμενη κοινή αξιολόγηση. Πολύ σημαντικό το έργο και μάλιστα φάνηκε και στην τελευταία μας συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόντες όλοι οι πρέσβεις των κρατών μελών. Αυτό πραγματικά ήταν πρωτοφανές στο τέλος, την τελευταία μέρα μιας τέτοιας αντιπροσωπείας. Και έδωσα το παρόν τόσοι ε, πρέσβεις, γιατί ήθελαν ακριβώς να ενημερωθούν για τα επιμέρους ζητήματα, τις σχέσεις μας με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα επισκεφτήκαμε και το Λευκό Οίκο. Και είχαμε κάποιον, κάποια συνομιλήτρια που μπορέσαμε έστω και μάλιστα σε αρκετά υψηλό επίπεδο να συζητήσουμε ζητήματα της ιδιωτικότητας και είπαμε ότι να κάνουμε κάτι καλύτερο από το είναι απλώς ένας ασφαλής λιμένας και ε, εκφράσαμε την ελπίδα η μετάβαση να γίνει απρόσκοπτα. Και φυσικά μπράβο και στη Γραμματεία που για μία ακόμη φορά έκανε εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, μπράβο στη Γραμματεία μας. Αλλά μπράβο και στα μέλη της Επιτροπής που συνέβαλαν στην επιτυχία της αποστολής. Θα βάλω τελεία εδώ γιατί θα μπορούσα να μιλάω επί μακρόν. Δύο μέλη έχουν μείνει από την αποστολή, κυρία Μπεσέλη, και κυρία Τσινίτση, δεν ξέρω αν θέλουν σύντομα να πούν δύο λόγια. Η κυρία Κινίτσι. Ναι, ευχαριστώ, Κλοντ. Θα ήθελα και εγώ να ε, παρέμβω. Έχει περάσει και η ώρα και ούτως ή άλλως και μεταξύ μας είμαστε. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα για την αποστολή μας. Καταρχάς να ευχαριστήσω εσένα Κλοντ, διότι πραγματικά έκανες ε, συντονισμό και κατήφθηνε εντό εισαγωγικών όλη την αποστολή και την ομάδα. Ήμασταν μια ομάδα συναδέλφων που πραγματικά ε, ε, αντιμετωπίσαμε ενωμένοι το θέμα αυτό και εσείς ε, αυτός που έδωσε το βήμα για να συνεργαστούμε τόσο καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη τη γραμματεία που είναι εδώ παρούσα και όλους εκείνους που πραγματικά εργάστηκαν ώστε η αποστολή μας να μπορέσει να επιτύχει το στόχο της. Δηλαδή να γίνουν κάποιες ε, πολύ σημαντικές συναντήσεις υψηλού επίπεδου, το ανέφερες και εσύ, σε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας που εργαζόμαστε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και κατά την άποψή μου όλες αυτές οι συναντήσεις ήταν θετικές υπό την έννοια ότι επρόκειται και για συναντήσεις οι οποίες όντως ήταν ε, σε μια μεταβατική περίοδο, όχι τόσο για πολιτικό λόγους, αλλά γιατί άλλαζαν γραφεία οι άνθρωποι εκεί. Και καταφέραμε να κάνουμε παρόλα αυτά συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου στα θέματα τα οποία μας παρουσίασες προηγουμένως. Πρέπει να πω ότι για μένα όλα αυτά ήταν και προσπάθησα να συμβάλλω και στην ε, αποστολή, ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά εγώ προσωπικά βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικό το θέμα τη αντιμετώπιση τη τρομοκρατία και επομένω τη συνεργασία και τη ανταλλαγή των πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατά την άποψή μου πολύ σημαντική ήταν και η δυνατότητα να μπορέσουμε να επισκεφτούμε και να συναντήσουμε ε, τους του ε, Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας, το National Counter-Terrorism Center. Και αυτό το οποίο προέκυψε από εμά ε, και είναι πολύ θετικό, ε, είναι η καλή συνεργασία μεταξύ αρχών των ΗΠΑ Πολιτειών και Europol, αλλά και όχι μόνο της Europol, αλλά και κρατών μελών. Και κατά την άποψή μου αυτό ήταν από τα πιο ε, σημαντικά ε, σημεία αυτής της αποστολής, διότι ε, φάνηκε σαφώς ότι υπάρχει διάθεση να συνεχιστεί αυτή η αδιαλλαγή των πληροφοριών, που είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του διεθνούς ε, τρομοκρατικού εγκλήματος. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα ήταν το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Διότι και εκεί ε, διαπιστώσαμε τι επιλογές έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες έχουν επιλέξει να αναθέσουν εξωτερικά το θέμα της αντιμετώπισης της ε, ριζοσπαστικοποίησης ε, σε επίπεδο ομοσπονδίας ε, για να μπορέσουν λοιπόν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε και εμείς υπόψη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, τη ριζοσπαστικοποίηση. Ένα τελευταίο και με αυτό ολοκληρώνω που ήταν ενδιαφέρον ήταν τα μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο και επομένως και η δυνατότητα να αφαιρείται περιεχόμενο το οποίο προτρέπει σε μίσος. Εδώ βλέπουμε ότι διαφέρει πολύ η κατάσταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, όπου η ελευθερία έκφρασης, ε, την οποία εγγυάται η πρώτη τροπολογία του συντάγματος, περιπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα. Ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα ε, και αυτούς που τελικά είναι αρμόδιοι για να λάβουν ε, την τελική απόφαση για τη διαγραφή μηνυμάτων μίσους και ε, την ελπίδα που εξέφρασαν οι επιχειρήσεις να είναι οι αρχές οι οποίες αυτές θα αναλαμβάνουν την ευθύνη, ε, οι αρμόδιες αρχές, ε, καθορίζοντας ε, και πιο σαφή νομοθεσία. Προέκυψε λοιπόν και αυτή η διαφορά στην τοποθέτηση. Ολοκληρώνοντας να πω και πάλι ότι ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν και τη γραμματεία. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή και ε, για τις συναντήσεις αλλά και για τις γνώσεις που αποκομίσαμε από την όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω το, το προσωπικό μας. Βέβαια πέρασε πολύ καιρό, αλλά η συνάντηση με το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας ήταν πραγματικά υπόδειγμα πόσο άρτια οργανωμένοι ήμασταν. Και το ίδιο και εκείνοι. Και είχαμε πολύ υψηλόβαθμους εκπροσώπους και της Αμερικανικής Διοίκησης. Ε, πολύ ψηλότερα κλιμάκια από ό,τι συνήθως μας συνάντησαν. Και αυτό δείχνει σε τι οριμότητα έχουν φτάσει οι επαφές μας και η επικοινωνία μας με την Ουάσιγκτον. Η Τερέζα Μπεσερίλ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας να σε ευχαριστήσω, Κλοντ, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολες ε, τέτοιες αποστολές και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν ήταν εύκολη αποστολή ούτε για σένα, Κλοντ. Παρ' όλα αυτά έδωσε το παρόν, όπως είπε η Κατερίνα Κινίτση. Όχι μόνο έδωσε το παρόν, αλλά ήσουν και ιδιαίτερα δραστήριος και κατάφερες βουλευτές από διάφορες πολιτικές παρατάξεις με διαφορετική ιδεολογία σε μια χώρα από οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην πρωτεύουσα, τη Βάσιγκτον με τέτοια πολιτική πολυμορφία και σε τέτοια χρονική στιγμή, σε τέτοια συγκυρία με την ε, προεδρία του Πρόεδρου Τραμπ, παρόλα αυτά καταφέραμε εμείς να είμαστε συσπηρωμένοι, συμπαγείς, ενωμένοι και να εκπροσωπήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα όχι μόνο τι χώρε ε, των μελών της αντιπροσωπείας αλλά και τις χώρες που δεν είχαν μέλη στην αντιπροσωπεία αλλά που κρίναμε ότι έπρεπε να προστατεύσουμε όπως τις πέντε χώρες για τις οποίες απαιτείται βίζα για την είσοδο των υπηκών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πραγματικά ήταν κατάμεστο το πρόγραμμά μας και άρτια προετοιμασμένο και κάθε φορά όταν το κρίναμε σκόπιμο και εύστοχο επισημέναμε αυτό το ζήτημα τονίζοντας πόσο άδικο είναι κατά τη γνώμη μας και ζητήσαμε φυσικά την επίλυση με βάση την αμοιβαιότητα. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν τα θέματα του εμπορίου, όπως είπαν ο Κλώτ και η το θέμα του ασφαλούς λιμένα, και όλα τα ζητήματα που είχαμε σε προηγούμενες αποστολές μας στη Γόσικτον να πραγματευτεί. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι και ένα θέμα στο οποίο αφιερώνω τον περισσότερο χρόνο μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θέμα της τρομοκρατίας, το θέμα του κυβερνοεγκλήματος. Εκεί συναντηθήκαμε με επιχειρήσεις που ασχολούνται με την προστασία από το κυβερνοέγκλημα. Και ένα σημαντικό τμήμα της αποστολής ήταν η συνάντησή μας με εκπροσώπους των θυμάτων και ε, όχι τόσο με εκπροσώπους των θυμάτων, αλλά ε, εκπροσώπους κυβέρνησης που ασχολούνται με τα θύματα και από το Κογκρέσο και ανταλλάξαμε βέλτιστες πρακτικές. Επίσης συναντηθήκαμε με πολιτικούς, με γερουσιαστές, με την εκπροσώπους κυβέρνησης, πρέσβης. Πραγματικά επαναλαμβάνω άρτια οργανωμένη αποστολή, υπερπλήρες πρόγραμμα. Εμένα με άγγιξε ιδιαίτερη επαφή με τα θύματα, αλλά και με το Κέντρο Αντιτρομοκρατίας. Πολύ σημαντική η συνάντηση με το Κέντρο NCTC. Και μάλιστα ήταν πολύ ειλικρινή και άμεση η ανταλλαγή απόψεων και ήταν και πολύ καλές εξηγήσεις που μας έδωσαν. Αλλά και εμείς ήμασταν πολύ κατατοπισμένοι γιατί οι περισσότεροι ήμασταν εξοικειωμένοι με το θέμα και είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ε, γνωρίζαμε τα πράγματα εις βάθος. Δεν πήγαμε στην Αμερική μόνο για, για τουρισμό. Είχαμε κάνει μεγάλη προεργασία. Και θεωρώ ότι προασπίσαμε πολύ επάξια τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευχαριστώ θερμά τον Κλοντ, γιατί παρά τη θλίψη του και τη δύσκολη στιγμή που βίωνε προσωπικά, νομίζω τελικά τον βοήθησε αυτή η συμμετοχή του, το ότι τον περιβάλαμε με τέτοια στοργή και ένιωσε καλά και πέρασε έτσι αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή που ζούσε. Πάντως ήταν πολύ επιτυχημένη αυτή η αποστολή και μπράβο μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Η Λίμπε πηγαίνει τώρα στην Ουάσιγκτον ε, και θα αντιμετωπίζετε με πολύ περισσότερο σεβασμό. Τα προγράμματα είναι αναλυτικά, ε, πολύ καλή οργάνωση. Θα ήθελα να καταγράψεις ε, στα πρακτικά τις ευχαριστίες μου προς την γραμματεία. Και επειδή ούτε ή μεταδίδεται στο διαδίκτυο, θα το ακούσουν κάποιοι. Ο Χωσή Μανουέλ είναι εδώ, ο Μάικλ, όλο το προσωπικό μα. Θέλω να το ευχαριστήσω για την δουλειά που κάνει. Ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμα και με τον Έπλο και τους άλλους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκα ήταν κάτι πολύ θετικό. Και τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, το προσωπικό χαμογελά, ναι. Και με το προσωπικό πέρασαμε πολύ ωραία. Αλλά πιστεύω ότι ε, πραγματικά ε, υπερβήκαμε αν θέλετε και το ανάστημά μας ε, στην ΟΑΣΚΟ. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και σας ευχαριστώ και τις δύο συναδέλφους βουλευτές. Έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Η αντιπροσωπεία μας στην Αλλη του τώρα στο Τόκιο πολύ σύντομα. Είναι κανείς εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ, μόνο εγώ από όσους ήταν στην ε, επίσκεψη αυτό και άρα τι να σας πω, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αποτελεσματικά οργανώθηκε αυτή η επίσκεψη. Εστιάσαμε κυρίως ε, ε, στην απόφαση περί καταλληλότητας, adequacy, σε σχέση ε, με την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία και αυτό ήταν το βασικό κομμάτι που μας απασχόλησε, όπως επίσης και η κυβερνασφάλεια. Πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Καλύψαμε τη συμφωνία κατάλληλα που ήταν το βασικό, αλλά τα κυβερνο, περί κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Εξαιρετική συνάντηση, εξαιρετική. Αλλά το επίκεντρο ήταν ότι αν θέλουμε να ολοκληρωθούν αυτές οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις που σημαίνει ότι τα πρότυπα μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να εναρμονιστούν. Τέλος πάντων υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Συναντήσαμε κάθε συνομιλητή δυνατό, από το Υπουργείο μέχρι ε, τους μεγάλους επιχειρηματικούς κλάδους, ε, τη Χιτάτσι, τη Σόνη. Ε, είδαμε επίσης ε, τους ομοτήμους, δηλαδή τους ομολόγους μας από τις αρχές προστασίας δεδομένων και Πραγματικά ενθουσιάστηκα με το αποτέλεσμα και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Λίμπε αλλά και τη Γραμματεία για την εξαιρετική αυτή επίσκεψη. Είναι προνόμιο να είμαι μέλος της Λίμπε και να κάνω αυτά που κάνω. Νομίζω ότι και οι Ιάπωνες μας ε, φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, γιατί και αυτοί θεωρούν τα ζητήματα αυτά σημαντικά, δηλαδή την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των εμπορικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. συμμετείχαν και αυτοί σε συζητήσεις που και για μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συμμετείχατε σε αυτήν την αποστολή. Ο Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ δεν είναι τώρα εδώ βέβαια, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ, ιδίως με τις γνώσεις που έχει. Βέβαια όλοι, όλα τα μέλη της ομάδας. Ήταν πολύ καλή η σύνθεση ομάδας, η Νάταλη και όλοι οι άλλοι η Μπάρμπαρα, η Νάταλη, ο Μάικλ. Πάρα πολύ καλή αντιπροσωπεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους και πάλι στη γραμματεία. Ήταν προνόμιο να είμαι στην αντιπροσωπεία αυτή. Αυτά λοιπόν. Επόμενο θέμα. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Τερέσα Κατερίνα, μόνο εσεί είστε εδώ. Αλλά επειδή μπορεί να μα ακούει κάποιο από το διαδίκτυο. Τα πιο ε, καλά, ε, οι, πιο, οι πιο καλοί συνάδελφοι είναι εδώ και δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερου για να του ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και το προσωπικό βέβαια. Δεν με ακούνε, ω συνήθω βέβαια. Μιλάνε μεταξύ του, αλλά δεν πειράζει. Πάντω εύχομαι σε όλου ε, ό,τι καλύτερο. Καλέ γιορτέ. Βέβαια θα τα πούμε και στο Στρασβούργο. Τι έχουμε κάτι τη Δευτέρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, έχουμε τον διάλογο ασφαλεία τη Δευτέρα, στην Επιτροπή Λίμπε. Δεν μπορώ να σας αποχαιρετήσω. Ποτέ δεν μπορεί κανεί να πει αντίο στην Επιτροπή Λίμπε. Ναι, έχουμε τον Επιτρόπο Κίνγκ. Έχουμε το διάλογο για την ασφάλεια. Άρα αφήστε τα ωρεβάρ και τα goodbye. Ξεχάστε τα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Στι 7. 7 το απόγευμα, ναι. Θα σας δω εκεί. Θα είναι μια πολύ καλή συνεδρίαση. Τα λέμε τη Δευτέρα λοιπόν για μια ακόμη συνεδρίαση Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αν υπάρχει κάποιος που δεν θα δώσω στρασβό από το προσωπικό, ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλές διακοπές.